Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, έχετε συνεδρίαση. Δεν θέλω να σας πω ότι μόλις ολοκληρώσαμε τη συνεδρίαση των συντονιστών μας, πριν από το μεσημέρι θα πάρετε τα αποτελέσματα της συνεδρίασης αυτής και σας παρακαλώ να τα έχετε διαβάσει μέχρι τις 3 το απόγευμα για να μπορέσουμε να τα εγκρίνουμε. Περνάμε το σημαντικό σημείο της σημερινής διάταξη. το διαδίκτυο είναι εκπαιδευτικό εργαλείο για την πολιτική κατανόηση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι ξέρουμε όλοι ότι οι τεχνολογίες ενημέρωση και ε, πληροφορική άλλαξαν τον κόσμο. Μεταξύ αυτών και το πώς μαθαίνουμε. Σήμερα με ένα, πατάμε ένα κουμπί και έχουμε μια πληθώρα πληροφοριών που μπορεί να επιλέξουμε. Έχει επίδραση στην άποψη των συμπολιτών μας, της κοινωνίας μας και υπάρχουν νέες άγουσες εκμάθησης. Αυτό τι σημαίνει για τη μελλοντική μα εργασία στον τομέα των πολιτισμικών Έχουμε το 167.4 στη συνθήκη τη Λισαβόνας. Δηλαδή σε όλους τους τομείς της πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το θέμα το πολιτισμικό. Έχουμε την ε, σύμβαση της UNESCO που, χρησιμοποίησαμε, που συζητήσαμε πολύ την περισμένη εβδομάδα και είχαμε και μία ακρόαση πάνω σε αυτή. Σύμβαση για Αποβολισμική Ποικιλομορφία και θα πρέπει λέω να προσπαθήσουμε όλοι να έχουν τις διαπολιτισμικών μεθόδων εκμάθησης και να συμμετέχουν σε έναν διαπολιτισμικό διάλογο. Θα πρέπει το υλικό που είναι στο διαδίκτυο να αντικατοπτρίζει τους διάφορους πολιτισμούς μπορεί να θα πρέπει να έχει κανένας ικανότητες για να το εκμεταλλευτεί όμως διάφορες δυνατότητες γλωσσών, κατανόηση των χρηστών για να μπορούν να χρησιμοποιούν τα διάφορα μέσα σωστά πριν από 15 χρόνια, 15 ε, μέρες ή στο Στρασβούργο μάλλον, υιοθετήσαμε το Ευρωπαϊάνα, που είναι ένα βήμα προς την ψηφιακή ε, μορφή του πολιτισμικών μας ε, κληρονομικών στοιχείων. Θα παράσουμε τώρα στην εξέταση αυτού του θέματος, για τους έχουμε επικρονομώσει τον κύριο Ιωάννη Στεγκρούτερ από το ε, Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λέβεν, τον κύριο Άντρη Ράση, από το Φόρουμ της Προσωπικής Δημοκρατίας. Μετά έχουμε την καθηγήτρια κυρία Βέρενα Βίντεμαν, που την ξέρουμε από πολλές ακροάσεις για ραδιο... τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και τον κύριο Ζωνζουέλ Τζενερή που είναι ιστορικός ονομάζεται ως πρόεδρος της Γαλλικής Εθνικής Βιβλιοθήκης και πρόεδρος της Partner. Προβλέπουμε να οργανώσουμε τον κρόσιο ως εξής. Θα έχουμε δύο γύρους των παρουσιάσεων των επιρρογνώμων. Πρώτο, The Cruiter ραστάι ο καθένας από 10 λεπτά. Θα συζητήσουμε μετά αυτά που θα μας πούνε. Μετά οι δύο επόμενοι μελτές, βίντεο Genene, με την ίδια διαδικασία και θα ήθελα να παρακαλώ στους αδέρφους ε, τις παρεμβάσεις να τις χρησιμοποιήσουν για την υποβολή ερωτήσεων πραγματικά για να μπορούμε να έχουμε ένα απτό αποτέλεσμα. Δεν θα πρέπει ο καθένα να κάνει μια δήλωση, α πούμε, και κατά σύνομες σύνομε παρεμβάσει για να μπορούν οι στην άλλη να πάρουν το λόγο. Έω το τέλο θα ακούσουμε σχόλια τη Κομισιόν και τη Ισπανική Προεδρία. Τώρα, όπως ξέρετε, περνάει στο web stream η συνεδρίαση αυτή. Πρέπει να σας το πω αυτό. Και σας παρακαλώ να κλείνετε τα μικρόφωνα σας μετά που θα έχετε μιλήσει. Αυτά. Θα ήθελα τώρα να χαιρετήσω και εξ τη της Κομισιόν τον κύριο Ματέο Τσαχέτη Γενική Διεύθυνση Παιδεία και Πολιτισμού και την Νέτα Τουλτούρ από την ε, Γενική Διευθύνσο και τον κύριο Χαβιέ Κοσάλε Ζέγκα και την κυρία Κοντελούπη Μελτουόζα από την Ισπανική Προεδρία. Αρχίζουμε τώρα την ακρόαση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γιωάννη Στεκρότερ από το Πανεπιστήμιο του Λέβεν. Παρακαλώ. You have the floor. Push the μου φαίνεται ότι βρήκα το κουμπί, λοιπόν. Θα ήθελα να μιλήσω σύντομα για την πλασματική κινητικότητα που είναι μια έννοια που χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιό μας για να στηρίξει τη διεθνή παιδεία μέσω της ηλεκτρονικής το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβένης είναι περίπου απέχει 30 λεπτά από εδώ. Και έχουμε όλες τις έδρες εκτός από την κτηνιατρική. Έχουμε 30.000 φοιτητά και φοιτητρία. Και συνδεόμαστε με άλλα 13 πανεπιστήμια. Έτσι έχουμε πρόσβαση σε περίπου 85.000 φοιτητές. Ιδρυθήκαμε το 1425 και είμαστε από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Οι νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες είναι μια έδρα που χρησιμοποιείται στο πανεπιστήμιό μας για, όπως λέει ο τίτλος, τη ηλεκτρονική εκμάθηση. Οργανώνουμε ειδικά μαθήματα και τμήματα ανάλογα με τις ανάγκες των φοιτητών. Εγώ ονομάζομαι Policy Advisor εκεί μέσα. Θα ήθελα τώρα να σας μιλήσω για το πώς εννοούμε τη διεθνοποίηση και παγκοσμιοποίηση καθώς και την έννοια της πλασματικής κινητικότητας. Ε, βασικά υπάρχουν πολλοί ορισμοί για την διεθνή παιδεία ή εκπαίδευση ή την διεθνοποίηση της εκπαίδευσης. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε αυτό καθώς έχει σημειωθεί και η παγκοσμιοποίηση. Καταρχάς υπάρχουν προγράμματα που μπορεί να χρηματοδοτούνται από την Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς και σε δεύτερο επίπεδο υπάρχει ένας οργανισμός, μία λέσχη πολλών πανεπιστημίων που εφαρμόζουν προγράμματα διεθνούς εκπαίδευσης επιτόπου. Δηλαδή οργανώνουν δραστηριότητες και εκδηλώσεις από άλλα πανεπιστήμια που δεν χωρίς να έρχονται οι εκπρόσωποι τους επιτόπου. Το κυριότερο παράδειγμα είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιεί η Λουβένη για να προσπαθήσει να διεθνοποιήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Έχει γίνει μια μελέτη όπου αναγνωρίστηκαν 8-9 τρόποι διεθνοποίησης των εκπαιδευτικών πανεπιστημιακών προγραμμάτων. Κυρίως για εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες. Η διεθνοποίηση της παιδείας λοιπόν σημαίνει παρακολούθηση προγραμμάτων σε διάφορα πανεπιστήμια είτε με μετακίνηση και ανταλλαγές είτε επιτόπου με τηλεδιασκέψεις. Νομίζουμε ότι η διεθνοποίηση αυτή συνδέεται με την πολιτισμική αλληλοκατανόηση διότι όταν κανείς ταξιδεύει βλέπει διαφορετικούς πολιτισμούς και καταλαβαίνει ότι μαθαίνει για τις πολιτισμικές διαφορές και έτσι είναι σε θέση να κατανοήσει καλύτερα τον πολιτισμό των άλλων. Αυτός βέβαια δεν είναι ο μόνος στόχος της διεθνούς εκπαίδευσης, μόνο. Κύριος στόχος, αρχικά τουλάχιστον, ήταν να ανταλλάξουν ακαδημαϊκές εμπειρίες οι φοιτητές και φοιτήτριες να επισκεφθούν ή να έχουν πρόσβαση σε ακαδημαϊκά προγράμματα από διαφορετικές χώρες από τη δική τους. Η διαπολιτισμική κατανόηση λοιπόν είναι κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί, αλλά βασικά είναι γνώση και δεξιότης για την πραγματικότητα άλλων πολιτισμών. Γι' αυτό βέβαια απαιτείται και η απαραίτητη περιέργεια και ενδιαφέρον. Δικό μας καθήκον εδώ είναι πώς να βοηθήσουμε τους καθηγητές να χρησιμοποιήσουν έννοιες όπως την πλασματική κινητικότητα για να διευκολυνθούν οι διεθνείς συνεργασίες στα πλαίσια της εδίας. Και επαναλαμβάνω ότι το θέμα δεν αφορά μόνο την εκπαίδευση καθεαυτήν αλλά και την έρευνα. δεν είναι τελείως πλασματική εμπειρία, μπορεί να σημαίνει και κάποια σωματική ανταλλαγή, φυσική ή την εκδήλωση σε διαφορετικούς τόπους διαφόρων γεγονότων. Την ονομάζουμε συνεργατική εκπαίδευση γιατί με την τεχνολογία του ίντερνετ μπορούμε να προσελκύσουμε πολύ κόσμο. Δεν πρόκειται απλώς για παθητική κατανάλωση πολιτισμικών αγαθών όπως βίντεο, αλλά υπάρχει και διάλογος και πρέπει να υπάρχει διάλογος και διάδραση. Ένα από τα κύρια θέματα που μας απασχολεί είναι η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας του ίντερνετ για να διοργανωθούν διεθνείς εκδηλώσεις με τον ίδιο βαθμό έντασης που θα είχαν και αν ήταν φυσικά παρόντες οι συμμετέχοντες όλοι. Είναι βέβαιο ότι αν θέλει κανείς να βιώσει πλήρως έναν άλλο πολιτισμό δεν μπορεί να το κάνει 100% μέσω της τεχνολογίας αλλά μπορεί να διευκολύνει η τεχνολογία αυτή περισσότερη πληροφόρηση και γνώση όπως ξένων γλωσσών ή διαφορετικών αξιών και θέσεων. Δεν μπορώ να πω ότι είναι το ίδιο με την σωματική εμπειρία. Διοργανώνουμε όπως σας είπα εργαστήρια, σεμινάρια διεθνώς χωρίς να χρειάζεται πάντοτε να μετακινηθούμε αλλά χρησιμοποιώντας τη τηλεδιάσκεψη και άλλα μέσα με το ίντερνετ για να συναντήσουμε κόσμο. Μπορούμε να τους δούμε, να τους μιλήσουμε, να δούμε τις εκφράσεις στο πρόσωπό τους. Και η τηλεδιάσκεψη είναι από τα κυριότερα εργαλεία που χρησιμοποιούμε γιατί η τεχνολογία αυτή οριμάζει όλο και περισσότερο και αυξάνεται η ποιότητα των τηλεδιασκέψεων. Έχουμε πλήρη οπτική επαφή με τους συνομιλητές, καλύτερο ήχο και οι ανταλλαγές που μέχρι τώρα ήταν κυρίως με βάση κείμενα τώρα είναι και οπτικές. Μερικά παραδείγματα για να τελειώσω. Πρώτον, σε μια σειρά γλωσσικών μαθημάτων χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο που χρηματοδοτήθηκε από την Κομισιόν όπου κάναμε, οργανώσαμε δικτυακές διασκέψεις όπου μπορούν να συνομιλήσουν οι φοιτητές με ένα πανεπιστήμιο του ΙΤΑΒ και όχι μόνο να συνομιλήσουν αλλά να αξιολογήσουν και όλα την εμπειρία τους να δούμε και εμείς πόσο καλά εκφράστηκαν στην ξένη γλώσσα και να δημιουργηθεί έτσι ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αξιολόγησης. Δημιουργήσαμε μία δωρεάν δικτυακή υπηρεσία όπου όσοι μαθαίνουν ξένες γλώσσες είναι σε θέση να συνομιλήσουν με ανθρώπους που μιλούν μια άλλη γλώσσα ας πούμε ένας Ολλανδόφωνος να συνομιλήσει με γαλοφόνους. Χρησιμοποιήσαμε την ιδέα αυτή που προϋπήρχε και σε ακαδημαϊκό επίπεδο και κάναμε και την τελική αξιολόγηση. Είναι εδώ αυτό ένα παράδειγμα χρήσης διαπολιτισμικών ανταλλαγών. Κάποιος μιλάει χωρίς μικρόφωνο, η κυρία Πακ μάλλον. Με αυτή την υπηρεσία το web surf δηλαδή μάθαμε ότι παρά την επιτυχία της εμπειρίας πολλοί ήθελαν να την παρατείνουν και σε άλλους τομείς. Όχι μόνο στην εκμάθηση γλωσσών αλλά ήθελαν να αξιολογηθούν και στο κατά πόσον ήταν ικανοί και αποτελεσματικοί στη χρήση της ξένης γλώσσας. Αποφασίσαμε λοιπόν το εργαλείο αυτό να το επεκτείνουμε και τώρα το μελετάμε. Χρησιμοποιούμε δε την κλίμακα ίνκα που είναι ένα από τα προγράμματα του Λεωνάρδου από το 2004 που αξιολογεί κατά πόσον κανείς μπορεί να εκφραστεί σε μια ξένη γλώσσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Άλλο παράδειγμα που δεν είναι καθαρά δικό μας αλλά του Imperial College του Λονδίνου είναι ένα πρόγραμμα διεθνών επιχειρήσεων όπου φοιτητές ε, οικονομικών μαθημάτων ή διεύθυνση επιχειρήσεων πρέπει να διευθύνουν μία πλασματική εταιρεία σε όλα τους τα επίπεδα και μάλιστα πολυγλωσσικά. και διάφορα σενάρια μπορούν να παιχτούν με αυτό το εργαλείο. Και ε, τα σενάρια που ήδη υπάρχουν αφορούν μεταξύ άλλων ας πούμε εργασιακές, εργασιακά προβλήματα και διαφορές. Επίσης στο Πανεπιστήμιο της Λουβένης εδώ και δέκα χρόνια υπάρχει ένα μάθημα που λέγεται Film and Literature και εδώ διοργανώνονται κοινά μαθήματα με τηλεδιάσκεψη όπου δεν βλέπουμε μόνο τους καθηγητές να διδάσκουν αλλά οργανώνονται και συζητήσεις μεταξύ φοιτητών και φοιτητριών. τα θέματα επιλέγονται από κοινού από όλους τους συμμετέχοντες και οι φοιτητές μπορούν να συζητήσουν το εύρος του θέματος μεταξύ τους και να το συγκρίνουν με μαθήματα ανάλογα σε άλλες χώρες και πανεπιστήμια. οι φοιτητέ και οι φοιτήτριε μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δική τους γλώσσα ή μια ξένη γλώσσα κατ' επιλογή. Και ελπίζουμε ότι με αυτή τη συνεργασία θα ελκύσουμε τους φοιτητά και φοιτητρίας να ενδιαφερθούν και για τον πολιτισμό της άλλης χώρας. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ως λεπτομέρειες γιατί είναι τμήμα της μαθησιακής εμπειρίας. Ας παραλείψω τώρα μερικά για να σας αναφέρω μόνο ότι χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική τεχνολογία κυρίως για την διοργάνωση φοιτητικών ανταλλαγών πριν πάει κανείς στην άλλη χώρα, για την οργάνωση ήδη της ανταλλαγής. Υπάρχει το πρόγραμμα «Πλασματικός φίλος» όπου φοιτητές συναντιούνται στο διαδίκτυο και μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες και στην καλύτερη περίπτωση να δημιουργήσουν και φιλίες. Και δημιουργούνται έτσι και δίκτυα των αποφοιτησάντων. Και άλλοι δημιουργούν δικά τους δίκτυα μετά. Ήταν μεγάλη επιτυχία στην αρχή δεν το είχαμε συμπεριλάβει μέσα στο θέμα των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, αλλά τώρα βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για την προετοιμασία των πολιτιστικών ανταλλαγών. Και τώρα, αν έχετε απορίες, με τα χαράς να σας τις λύσω. Ελπίζουμε να αναγνωριστεί και να υποστηριχθεί και χρηματικά η εμπειρία αυτή, όχι μόνο από τον έρασμο αλλά και από άλλα προγράμματα. Μέχρι το 2020 θέλουμε να φτάσουμε σε κάποιο προκαθορισμένο επίπεδο ποσοστιαίο αριθμού φοιτητών που ασχολούνται με τέτοιου είδους ανταλλαγές γιατί έχει αποδειχτεί ότι εμπλουτίζει την εμπειρία τους. Γι' αυτό βέβαια χρειάζεται και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και υλικό. Αλλά δεν είναι αυτό το κυριότερο. Δεν χρειάζονται τεράστια ποσά, αλλά κάποια οπωσδήποτε. Η πρασματική κινητικότητα είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό για μας. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα ο κύριος Ρασιέ. Ορίστε κύριε μου. Good morning, everyone, and, uh... Καλημέρα σε όλους και σας ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Θα ήθελα να πω ότι η διακοπή που είδαμε πριν από πέντε λεπτά ήταν ακριβώς αυτό που κάνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προσπαθούν να διακόψουν τη συζήτηση για τα νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ελπίζω να μην με διακόψετε και εμένα με τον ίδιο τρόπο. Το διαδίκτυο είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα του κόσμου ήδη για να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και όλοι πλέον είμαστε ένα σύνδεμο μακριά ο ένας από τον άλλον. Και παρά το γεγονός ότι σήμερα κοιτάμε να δούμε τι μπορούν να κάνουν κυβερνήσεις, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όλοι κολυμπάμε στα ίδια βαθιά νερά της ε, τεχνολογίας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όλοι ξέρουμε και όλοι διαβάσαμε πως η εκστρατεία του Ομπάμα το 2008 χρησιμοποίησε το διαδίκτυο με επιτυχία για να προωθήσει την υποψηφιότητά του. Ως φοιτητή πολιτικής και τεχνολογίας δεν είχα αντιληφθεί πόσο είχε αλλάξει ο κόσμος μέχρι που επισκέφθηκα τον πατέρα μου ένα απόγευμα διότι μου τηλεφώνησε, μου ζήτησε να πάω στο σπίτι του να τον βοηθήσω με το email του. Ο πατέρα μου δεν είναι και πολύ πολιτικοποιημένο άτομο. Δεν θα πήγαινε ποτέ σε ε, διαδήλωση, ούτε θα σήκωνε κάποιο πλακάτι για υποψήφιο, ούτε θα τηλεφωνούσε στους φίλους του να τους πει ποιο να ψηφίσουν. Αλλά αν βρεθεί σε ένα δείπνο ή με κάποιους φίλους σε ένα εστιατόριο ή στο σπίτι ε, και τύχει να συζητηθεί πολιτική, θα πει την άποψή του. Ο πατέρας μου είναι 83 ετών. Κατανοείται λοιπόν ότι ψήφιζε στι Ηνωμένε Πολιτείε από τα 50 του και λίγο πολύ σε όλε τι εκλογικέ αναμετρήσεις αυτό έκανε και αυτή ήταν η σχέση του με την πολιτική. Εκείνο το απόγευμα όμω προσπαθούσα να το βοηθήσω με το email του γιατί δεν ήξερε πώ μπορεί να στείλει περισσότερα μηνύματα ταυτόχρονα. Και όταν τον βοήθησα είδα τι έγραφε στο email και ήταν ένα σύνδεσμο για να δει ένα βίντεο του Μπάρακ Ομπάμα στο YouTube. Και αυτό που έγραφε ήταν απλώ δείτε το. Αυτό που κατάλαβα ήταν ότι ο πατέρας μου μιλούσε με τους ίδιους 50 ανθρώπους με τους οποίους ε, συναντιόταν κοινωνικά στο ίδιο εξάμεινο σε ένα απόγευμα με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού τεχνίου. Ο πατέρας μου είχε γίνει λοιπόν ένα πολιτικό πρόσωπο του 21ου αιώνα και δεν το είχε καν αντιληφθεί. για να έχετε μια εικόνα του τι ακριβώς σημαίνει αυτό για όλο τον πληθυσμό των ΗΠΑ, στις προεδρικές εκλογές του 2008 είχαμε 1,5 δισεκατομμύριο ε, βίντεο ε, online, τα οποία παρουσίαζαν είτε τον Μπάρακ Ομπάμα είτε ναι. το Μακέιν. Και από αυτά τα 1,5 δις ε, βίντεο, 1,35 δις ήταν βίντεο τα οποία είχαν ετοιμάσει οι ίδιοι οι πολίτες. Δεν ήταν τμήμα της προεκλογικής εκστρατείας. Είναι σαφές λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε πλέον κατά νου ότι οι άνθρωποι θα φτιάχνουν βίντεο και θα κάνουν πράγματα για να επικοινωνούν με τους άλλους πολύ πιο γρήγορα από τις κυβερνήσεις και δεν θα περιμένουν τις κυβερνήσεις να το κάνουν. Επίσης θα αναπτύξουν μια κοινή γλώσσα για να κατανοούν ένα τον άλλον, αντί να βασίζονται ο ένας στη γλώσσα του άλλου. Επίσης θα χρησιμοποιούν τα βίντεο ως εργαλεία και όχι το κείμενο πλέον, και εγώ έφτιαξα ένα καινούριο όρο που λέγεται βίντεραση, που σημαίνει ε, πόσες γνώσεις έχει κάποιος σε επίπεδο βίντεο. Φαντάζομαι ότι ο καθένας από εσά εδώ στην αίθουσα είναι μισοαγράμματος σε θέματα βίντεο, γιατί όλοι μπορούμε να ε, δούμε βίντεο, τα βλέπουμε στην τηλεόραση, στο DVD και online στο ίντερνετ, χωρίς πρόβλημα. Αλλά αν μας ζητήσετε να ετοιμάσουμε ένα βίντεο, ε, πολύ λιγότεροι από τους όσους βρίσκονται στην αίθουσα μπορούν να ετοιμάσουν ένα βιντεάκι. Δύσκολα. Και αυτούς τους ανθρώπους εγώ τους αποκαλώ βίντερα, γιατί έχουν αυτή τη βίντεραση. Γνωρίζουν πώς να φτιάχνουν βίντεο και δεν χρησιμοποιούν το κείμενο για την επικοινωνία, αλλά χρησιμοποιούν το βίντεο. in relation to the European Union.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 Λοιπόν, τι σχέση τώρα έχει αυτό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οργάνωσή μου, η Personal Democracy Forum, εξετάζει πώ ε, μπορεί η τεχνολογία να αλλάξει την πολιτική και την κυβέρνηση και την κοινωνία στι ΗΠΑ Πολιτείες τα τελευταία 7 χρόνια. Πέρσι ε, έγινε και το Ευρωπαϊκό Τμήμα στη Βαρκελόνη και, εξετάσαμε να εξετάζουμε, ε, και αρχίσαμε να εξετάσουμε τα θέματα Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε μια διμερίδα και προσπαθούσαμε να απαντήσουμε ερωτήματα για το πώ μπορεί η νέα τεχνολογία να έχει επιπτώσει στο σύστημα της Ευρωπαϊκής και πώς μπορεί να επισέλθει σε μια ευρύτερη πανευρωπαϊκή συζήτηση. Και εδώ είχαμε ένα φάσμα νέων ερωτήσεων και ελάχιστων απαντήσεων. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία είναι πλέον υπερεθνικά ε, και δημιουργούνται με πολύ φυσικό τρόπο και δημιουργούνται σύνδεσμοι πέραν των ε, ε, συνόρων των κρατών. Αυτό περιλαμβάνει και τη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, την ενίσχυση της διαφάνεια, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και φυσικά οι ελευθερίε στο διαδίκτυο. Υπάρχουν και κάποιες διαφορές, τις οποίες δεν μπορούμε να γεφυρώσουμε πολύ εύκολα. Ε, οι άνθρωποι ενδιαφέρονται να μάθουν πώς αλλάζει το διαδίκτυο την πολιτική στις ε, χώρες, αλλά αυτές οι αλλαγέ διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Στις πρόσφατες Βρετανικές εκλογές, για παράδειγμα, ε, είχαμε μια προεκλογική εκστρατεία μόνο τριών εβδομάδων και το διαδίκτυο είχε πολύ ελάχιστη επίπτωση σε σχέση με τα όσα συνέβησαν στις ΗΠΑ το 2008. Και επίσης ο κόσμος δεν μαθαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου, αλλά προσπαθούν να βρουν μια κοινή γλώσσα. Ο Ζερεμί Ζίμερμαν της La Quadrature du Net είπε ότι θα υπάρχει μια κοινή γλώσσα για την ε, πανευρωπαϊκή ε, συζήτηση ε, στο διαδίκτυο, μόνο όμως θα είναι τα αγγλικά. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα κοινό θέμα, προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε την διαδικτύα κυβέρνηση να λειτουργεί καλύτερα και πολλοί θεωρούν ότι μπορούμε να έχουμε ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή ε, κυβέρνηση 2, δηλαδή τη νέα εκδοχή. Εμείς έχουμε μια νέα ιδέα, το λέμε We Government και είναι ε, ένας χώρος στον οποίο οι άνθρωποι συλλέγουν στοιχεία ή από τις κυβερνήσεις ή συλλέγουν στοιχεία μεμονωμένα και δημιουργούν νέα φόρουμ υπηρεσιών και ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ των ώστε η ζωή τους και η κοινωνία των πολιτών να είναι πιο χρήσιμη και όλα αυτά γίνονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι τα κάνει η κυβέρνηση. Γι' αυτό ακριβώς σας ε, βρείτε τι ακριβώς σημαίνει ο όρος ε, open data, ανοιχτά δεδομένα και τι σημαίνει και δημόσια δεδομένα. Και επίσης, να σκεφτείτε ότι ο όρος δημόσιος σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να ψάξει κάποιος και να διαβάσει μέσω μιας μηχανής αναζήτησης ε, στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάτι καινούριο στον τρόπο με τον οποίο ορίζουμε τις δημόσιες πληροφορίες. Ένα στοιχείο ή μία πληροφορία σε ένα αρχείο ενός κυβερνητικού ε, φορέα δεν σημαίνει ότι είναι δημόσιο απαραίτητος. Υπάρχει και μία ακόμα κοινή γλώσσα την οποία μεταφέρει το διαδίκτυο και αυτό είναι χαλαρά τμήματα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί ισχυροί σύνδεσμοι και δεν είναι μόνο το HTML και οι υπερσύνδεσμοι, αλλά είναι και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε ταχύτατα να ανταλλάξουμε πληροφορίες. Τώρα, αν αυτό θα γίνει μέσω ενός θέματος στο Twitter ή από ε, τηλεδιασκέψεις ή από το Meetup Everywhere, που είναι πλατφόρμα που ε, κανονίζει συναντήσεις με ανθρώπους για να βρεθούν από εκεί και πέρα κάπου σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αλλά το βασικό θέμα που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι πώς μπορούμε να περάσουμε από την οικονομία της έλλειψης στην οικονομία της αυθονίας. Και η ταχύτητα είναι αστρονομική. Σε πέντε χρόνια εκτιμάται ότι όλη η ανθρωπότητα θα είναι διασυνδεδεμένη μέσω κινητών συσκευών και οι κινητές συσκευές που θα έχουν και θα έχουμε κατά χέρι, στο χέρι μας ε, θα κάνουν τα iPhone και τα BlackBerry που κρατάμε τώρα να φαίνονται σαν χαρτοφύλακες που είχαμε στα χέρια μας πριν από 20 χρόνια. Θα ήθελα τώρα να σταθώ στην ίδια την παιδεία και να σας εξηγήσω γιατί αυτή η ταχύτητα είναι τόσο σημαντική και γιατί το να αναπτύξουμε μια ισχυρή πολιτική για την κοινωνία της πληροφορίας ε, στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό. Πριν από 30 χρόνια ξεκίνησα μια μη κυβερνητοσκοπική οργάνωση στη Νέα Υόρκη που λεγόταν MAUS. Όταν ξεκινήσαμε το 1977, διαπιστώσαμε ότι οι τεχνολογίες πληροφορίας που χρησιμοποιούνταν στα δημόσια σχολεία ήταν ακριβώς οι ίδιες που είχαν και επιχειρήσεις. Δηλαδή είχαμε φαξ, ε, τηλέφωνα, ε, φωτοτυπικά μηχανήματα και ε, Υπολογιστέ ε, σε γραφείο που ήταν ουσιαστικά επεξεργαστές κειμένου και κανένας ε, σχεδόν δεν χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γιατί δεν υπήρχε. Τι συνέβη όμω σε 20 χρόνια, σε 13 συγγνώμη χρόνια. Σε 13 χρόνια κάθε επιχείρηση ανά τον κόσμο είναι συνδεδεμένοι και έχουμε δίκτυα τα οποία λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Αν αγοράσετε, για παράδειγμα, μία δερμάτινη θήκη για την φωτογραφική σας μηχανή από το αγαπημένο σας online μηχάνημα, με το που πατάτε το κλικ, ε, ε, το ταμείο το γνωρίζει, γιατί τόσο γρήγορα λειτουργεί το διαδίκτυο. Πού είμαστε όμως σε θέματα παιδείας. Τα σχολεία είναι ανοιχτά κατά μέσο όρο 20% ενός έτους οι κυβερνήσει ουσιαστικά έχουν το μονοπόλιο για να δίνουν, προσδίδουν παιδεία, εκπαίδευση, αλλά φανταστείτε τώρα οι οικογένειε ε, και οι κυδεμόνε να είναι συνδεδεμένες με τα παιδιά τους με τον ίδιο τρόπο που είναι επιχειρήσει. Οι φοιτητέ, οι μαθητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και η κοινωνία των πολιτών μπορεί να έχουν πρόσβαση στι ε, μεγαλύτερε, για παράδειγμα, βιβλιοθήκε του κόσμου, να μπορούν να έχουν ε, την εικόνα της δημοκρατίας του 21ου αιώνα που πηγαίνει πέραν των συνόρων και δημιουργεί ένα νέο όραμα για τη διακυβέρνηση της ανθρωπότητας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Φτάνουμε τώρα σε μια συζήτηση, ένα γέρο συζήτηση πάνω στις δύο αυτές ε, παρουσιάσεις. Ποιος θα ήθελε πρώτος το λόγο. Παρακαλώ. Μία ερώτηση στον δεύτερο μιλητή. Θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα όπου όλοι πρέπει να διδαχθούν και όχι μόνο μια ελίτ και όλοι πρέπει να πετύχουν. Και πρέπει να υπάρχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο θα στοχεύει στο μαθητή, ε, το οποίο διαφέρει από αυτό που είχαμε στο παρελθόν. Θεωρείτε ότι η εισαγωγή της τεχνολογίας και κυρίως του διαδικτύου προϋποθέτει ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο το οποίο θα διαφέρει από αυτό που είχαμε στο παρελθόν. Δηλαδή με νέα προγράμματα σπουδών, χωρίς ε, να κυριαρχεί η έδρα στην παλιά αίθουσα που θυμόμαστε ακόμα και από τα 1800, ίδιες είναι οι αίθουσες των σχολείων, και αν θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει όλο το εκπαιδευτικό σύστημα και όχι μόνο για λόγους τεχνολογίας και όχι γιατί έχουμε πλέον έναν εγγονικό κόσμο αλλά και γιατί πρέπει να δώσουμε πλέον έμφαση από τη διδασκαλία στην μάθηση. We are collecting uh, some, some questions. Okay? Please take note. Mr. Zver from Slovenia. Hvala lepa, predsednica. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ έχω μία ερώτηση προς τον κύριο Τικρόιτερ θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσον σήμερα ήδη οι φοιτητέ μπορούν να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο αυτό με μια ε, πνευματική κινητικότητα. Είναι δυνατόν δηλαδή να σπουδάσει κανένα στο πανεπιστήμιο χωρίς να είναι πραγματικά παρόν εκεί. Και δεύτερον, αυτό το πρότυπο μελέτης στο μέλλον θα αντικαταστήσει την πραγματική κινητικότητα των φοιτητών. Vielen Dank. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για... Ευχαριστώ για τόσο ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση για μια τόσο... ένα τόσο φουτουριστικό όραμα που θα γίνει στην πραγματικότητα. Οι, πληροφο... Οι πληροφορικής βέβαια δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την άμεση επαφή διδασκόντος και διδασκομένου. Γιατί αυτό νομίζω είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μόνο σε προσωπικές επαφές. Ε, έχω μια ερώτηση όμως που αφορά το εξής. Θεωρείτε ότι θα υπάρχει παντού στην Ευρώπη διαθέσιμο το διαδίκτυο ευρείας φάσης ε, και δεν θα υπάρχει πουθενά κανένα κενό. Μέσα στα πλαίσια αυτού του οράματος πιστεύετε ότι αυτά τα συστήματα ανταλλαγή φοιτητών, ανταλλαγή ε, μαθητών, ε, το να μάθει κανένας γλώσσε ή μάλλον οι φοιτητέ των νομική να μαθαίνουν ξένε γλώσσε. Αυτό συζητήσαμε τις προάλλες. Σήμερα οι φοιτητέ της νομικής δεν μπορούν να επικοινωνήσουν γιατί δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι, τέτοια σχέδια όπως το έρασμος θα μπορούσε να αντικαταστεί από ένα ηλεκτρονικό έρασμος δηλαδή. Αυτή η ανταλλαγή να γίνεται μέσα, στο διαδίκτυο. Mm. Ίσως χρειαζόμαστε ήδη πιλωτικά προγράμματα για κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ κύριε Νότουλα. Mulțumesc, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την εμπειρία των ε, επισκεπτών μας και να υποβάλω μια ερώτηση εν ώψη του ότι το ρυθμός ανάπτυξης τα τελευταία 10-15 χρόνια ήταν πάρα πολύ ψηλός, και επειδή οι προοπτικές που μας παρουσιάστηκαν επίκυνται πραγματικά να πραγματοποιηθούν, θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσον αυτή τη στιγμή Υπάρχει μία προοπτική για τις εξελίξεις τα επόμενα 50 με 100 χρόνια στον τομέα αυτό. Γιατί φαντάζομαι ότι θα διατηρηθεί ο ίδιος ρυθμός ανάπτυξης στην πληροφορική. Γιατί πραγματικά αυτός ο ρυθμός τα τελευταία 10 χρόνια ήταν καταπληκτικός και αναρωτιέται κανένας τι θα γίνει τα επόμενα 50 με 100 χρόνια αν συνεχίσουμε τον ίδιο ρυθμό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Πορτογαλία, κ. Καμπέλα. Ήταν πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσε αυτέ οι παρουσιάσει. Κάτι που έλεγε όμω. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες, αλλά να λάβουμε υπόψη μα και τι απειλές στην πολιτική, στην παιδεία. Θα πρέπει να μπορούμε να ελέγχουμε τον τομέα τη πληροφορική. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συστήσουμε. Και μετά μία ερώτηση προς τον ε, κύριο Ντουγκρότερ. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ανταλλαγή μεταξύ ε, φοιτητών και καθηγητών και διδασκόντων. Υπάρχουν ε, ίσως κάποιες ε, έρευνες που έχουν γίνει, ποιες είναι οι εμπειρίες που έχουν οι φοιτητές και οι καθηγητές στις ανταλλαγές μέσω διαδικτύου. Πρώτα σε ευχαριστώ. Θα ήθελα να πιστεύω την προσοχή στον που Μπορίσο ότι εδώ και πολλά χρόνια μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Κομένιους έχουμε ένα πρόγραμμα που λέγεται e-twinning, θαυμάσιο πρόγραμμα που ενώνει ε, ε τάξεις ε, σχολείων πέρα από τα σύνορα της Ένωσης. Είμαστε πάρα πολύ προχωρημένοι λοιπόν με αυτό το σύστημα Κομένιους που δεν είναι ένα σύστημα μονάχα άμεσης επαφή και ήμουν σε μια άλλη διάσκεψη σχετικά στη Σόφια πριν από κάποια χρόνια όπου συναντήθηκαν πάρα πολλά στάξη σχολείων με τους δασκάλους τους και είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανένας πώς αυτή η τεχνολογία ενώνει τους ανθρώπους, ενώνει τους μαθητές. Πώς εμπλουτίστηκε η ζωή τους με την επαφή αυτή και ας ήταν και πλασμική. Αυτό ήταν πραγματικά καταπληκτικό. Λοιπόν, δεν θα δώσω το λόγο τώρα στους εμπειρογνώμονες. Στον ε, κύριο Ράσια πρώτα. χωρίς μικρόφωνο και άνευ μικροφώνου. Μάλιστα. Οι ερωτήσεις σχετίζονται και με τους δύο μιλητές, αλλά θα φροντίσω να απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. η έννοια της ίδιας της παιδείας θα αλλάξει. Ιστορικά χαρακτηριζόταν από την σπάνιδα, την έλλειψη φοιτητών και φοιτητριών και εφήτη κανείς περιορισμένο χρόνο και έπρεπε να αποστηθίζει τη γνώση που του δίνανε και να είναι σε θέση μετά να επαναλάβει. Αλλά σε μια οικονομία όπου υπάρχει μεγάλος πλούτος πληροφόρησης η αποστήθηση δεν είναι απαραίτητο προσόν πια. Αλλά μάλλον ο τρόπος πλοήγησης του ανθρώπου στον κόσμο και αυτό απαιτεί κάποια τεχνολογική γνώση, ψηφιακή μάλιστα γνώση, για να είναι κανείς σε θέση να ψάξει και να ελέγξει την ποιότητα της πληροφόρησης χωρίς να εξαρτάται από τον καθηγητή ή την καθηγήτρια. Δεύτερον, που ρώτησε κάποιος Πολωνός εδώ. Οι καθηγητές δεν θα είναι πια καποκαθέδρας σοφή, αλλά θα είναι οδηγητές του μαθητή στην πλοήγηση που ανέφερα. Και ίσως να χρειαστεί και κάποιο γενικότερο παιδαγωγικό πλαίσιο και φυσικά ο καθηγητής θα πρέπει να κάνει και την αξιολόγηση. Την αξιολόγηση. Αλλά επαναλαμβάνω ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από την έννοια της σπάνιδος και να καταλάβουμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο που υπάρχει άφθονη πληροφόρηση και οι φοιτητέ και φοιτήτριε μόνοι τους θα διαλέξουν την παιδαγωγική τους κατεύθυνση και τους οδηγούς των. Τέλος, ε, η ταχύτητα αυξάνεται. αλλάζει το δεσοξυριβονουκλεϊκό μας οξύ κάθε 20 περίπου χρόνια. Και όσοι γνωρίζουν πώς χρησιμοποιείται το Twitter, ο κελαϊδιστής, στους νέους του μέλλοντος θα θεωρηθούν απαρχαιωμένοι και όσοι είναι κάτω των 25 ήδη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο μέλλον δεν θα χρειάζεται καν ήδη μάλλον δεν χρησιμοποιούν το email, αλλά τον κελαϊδιστή. Σας ευχαριστώ. Να πω και εγώ κάποια πράγματα. Το κατά πόσον θα αλλάξει το επίκεντρο της προσοχής μας και αν θα περάσουμε από τη διδασκαλία στη μάθηση, ε, συμφωνώ. Ναι, μεν εστιάζουμε περισσότερο στη μάθηση και τίθενται συνεχώ νέοι στόχοι, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και νέε τεχνολογίε, όπω για παράδειγμα τα μέσα κοινωνική δικτύωση στο διαδίκτυο έχουν κάποιε επιπτώσει. Δεν είναι μόνο ένα μέσο λοιπόν το διαδίκτυο, διαμορφώνει και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μάθηση. Και ναι, μεν η μάθηση έχει αλλάξει, όπως και ο Τζόρτ Σίμον στον Καναδά, στο Πανεπιστήμιο της Μπάσκα, λέει ναι, είναι διαφορετικά τα πράγματα γιατί λειτουργούν διαφορετικά οι νεφρόνες και οι συνδέσεις στον εγκεφαλό σας, αλλά αλλάζει και το, η εστίασή μας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα ως δάσκαλος θα πρέπει να βάλετε πλέον το μαθητή στο επίκεντρο, γιατί δεν μπορείτε να διδάσκετε τα, παρα... πράγματα με τον παραδοσιακό τρόπο, διότι πλέον έχουν αλλάξει τα εργαλεία. Πρέπει να είναι πιο συνεργατικό το μοντέλο και όσο περισσότερα εργαλεία χρησιμοποιείτε στην εμπειρία και οι μαθητές, εσεί ως δάσκαλο πρέπει να αλλάξετε το επίκεντρο, το σημείο που εστιάζετε και να εστιάσετε σε άλλα σημεία προσπαθούμε και εμείς να πείσουμε τους δασκάλους ότι πρέπει να ε, είναι πιο δυναμικά τα πράγματα και όλοι συνειδητοποιούμε ότι ε, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που μαθαίνουμε και η ε, εκπαίδευση πηγαίνει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση τρέχοντας, επομένως πρέπει να αλλάξουμε και εμείς. Mm. Τα τελευταία πέντε χρόνια το συζητούσαμε πάρα πολύ ε, ότι πρέπει να ακολουθούμε την τεχνολογία, αλλάζουν τα πράγματα ταχύτητα και βλέπουμε πόσα πράγματα πρέπει να αλλάξουν στην παιδαγωγική και πρέπει να ξανασχεδιάσουμε κάποια προγράμματα σπουδών και κάποια μαθήματα. Είμαι αισιόδοξο βέβαια και δεν πιστεύω ότι θα γίνουν τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα, τουλάχιστον όχι για τα παραδοσιακά πανεπιστήμια. Το κατά πόσον έχουμε δραστηριότητες ε, δικτυακής κινητικότητας, ναι, για κάποια μαθήματα έχουμε, ναι, αλλά από την άλλη είμαστε πανεπιστήμια, έχουμε ένα φυσικό χώρο στον οποίο συναντιόμαστε, αλλά προσεγγίζουμε και άλλους και υπάρχουν και διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που επεκτείνουμε. Συνεργαζόμαστε με ε, το ανοιχτό πανεπιστήμιο ε, των κάτω χωρών για να δημιουργήσουμε ομάδες οι οποίες θα μπορούσαν ίσως να έρθουν και να παρακολουθήσουν μαθήματα και να μπορούν να παρακολουθούν και κάποια πράγματα όμως μέσω διαδικτύου ε, ανα πάσα στιγμή. το βασικό θέμα για την εικονική κινητικότητα είναι να βρούμε πανεπιστήμια που έχουν αντίστοιχα προγράμματα και να ξεκινήσουν ανταλλαγέ φοιτητών μεταξύ των πανεπιστημίων. Ε, πρέπει να είμαστε και εμεί προετοιμασμένοι, αλλά πρέπει και τα άλλα πανεπιστήμια να είναι προετοιμασμένοι και χρειαζόμαστε δίκτυα για να γίνουν αυτά. Δεν είναι πολλά τα πανεπιστήμια που νιώθουν ότι πρέπει να είναι το περιεχόμενό τους όλο ανερτημένο στο διαδίκτυο, διότι δεν λειτουργούσαν έτσι τα συστήματα στο παρελθόν, αλλά υπάρχει και εικονική κινητικότητα και πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. το κατά πόσον θα πρέπει να υποκατασταθεί το ε, πανεπιστήμιο και η φυσική παρουσία με τα εικονικά μοντέλα, ε, διαφωνώ απολύτως. Πιστεύω ότι ναι, μεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και αυτά τα μοντέλα της πληροφορικής, αλλά ε, θα πρέπει να υπάρχει και η φυσική παρουσία κάποιου. και πρέπει στους φοιτητές που είναι παρόντες στο πανεπιστήμιο να δώσουμε και την εμπειρία του πανεπιστημίου. Ε, ναι μεν μαθαίνουμε πάρα πολλά από τη φυσική παρουσία, αλλά το γεγονός ότι μπορούμε να το εφαρμόσουμε και από το, ε, το φυσικό περιβάλλον στο εικονικό περιβάλλον είναι σημαντικό. Θεωρώ ότι πρέπει να συμπληρώνει το πακέτο. Το κατά πόσον θα πάνε τα πράγματα γρήγορα, νομίζω ότι απαντήθηκε η ερώτηση. Τα πάντα προχωρούν πάρα πολύ γρήγορα και οι φοιτητέ ήδη θα έχουν βρει τη λύση μόνοι του. Αν δεν του έρθει αυτό που ζητούν από τον καθηγητή, θα το βρούνε μόνοι του και θα πάρουν και το πτυχίο του γιατί αυτό του χρειάζεται. Και ήδη τη βλέπουμε αυτή τη δυναμική κίνηση. Οι φοιτητέ δεν έρχονται στα μαθήματα γιατί πολλέ φορέ μαθαίνουν πολύ περισσότερα έξω από την τάξη και δυστυχώ αυτό με φοβίζει και πρέπει να το έχουμε κατά νου. Τέλος, αν πρέπει να κάνουμε έρευνα για αυτά τα πλεονεκτήματα, απολύτως, αλλά αυτό είναι το τμήμα της έρευνας και της ε, τεχνολογίας της παιδείας, το κατά πόσον υπάρχει κάποια αξία για την ε, τεχνολογία και πρέπει να σχεδιάσουμε τη διδακτική. Η τεχνολογία είναι το μέσο, μπορεί να επηρεάσει, αλλά από εκεί και πέρα ε, το πώς θα σχεδιάσουμε κάτι για να έχουμε αποτελέσματα είναι αυτό που μας ενδιαφέρει δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία της πληροφορικής. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που είναι πανταχού παρούσα η τεχνολογία. Επομένως το θέμα είναι αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και απλώς να δεχτούμε ότι θα υπάρχει παντού η πληροφορική. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ αυτό που ο ε, Υπήρχαν πάντα τα εξαποστάσεις επιστήμια τα πανεπιστήμια που το έζησα εγώ, είχα ένα ασκούμενο που σπουδάζει έτσι, ε, έχει προστευτεί πάρα πολύ με τις νέες τεχνολογίες. Πολύ πιο απλό. Δεν χρειάζεται να στείλει κανένα τίποτα με το ταχυδρομείο, το στέλνει αμέσω. Μπορεί να συμμετάσχει σε βίντεο ε, διασκέψεις, ε, όλα αυτά υπάρχουν. Έχουμε ένα πρόβλημα γιατί μιλάμε για μαθητές που πρέπει να εισαχθούν σε αυτό τον κόσμο, να έχουν αυτά τα μέσα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι δάσκαλοι που πρέπει να τους ενημερώσουν δεν το έχουν ζήσει αυτό καθόλου. Δηλαδή μαθαίνουν ταυτόχρονα με τα παιδιά. Και αυτό είναι το πολύ δύσκολο. Και νομίζω ότι στα πανεπιστήμια είναι ιδιαίτερα άκαπτο. Το είδαμε στη διαδικασία Μπολόνια πόσο δύσκολο είναι να καταστήσουμε τους ε, καθηγητές σε θέση αυτό που εκπαιδεύανε προηγουμένως σε πέντε χρόνια να το μετατρέψουν έτσι ώστε να εκπαιδεύεται ο φοιτητής σε τρία χρόνια. Οι δυσκολίες είναι δηλαδή πολύ μεγαλύτερες στους διδάσκοντες και όχι στους φοιτητές και θα πρέπει να φροντίσουμε οι διδάσκοντες να έρθουν στο ε, ανώτερο επίπεδο. Όσον αφορά το νέο πρόγραμμα διαβίου μάθησης, ε, είπαμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα πρόγραμμα που ασχολείται με τους διδάσκοντες. Έχουμε για τους φοιτητές, για τους μαθητές, για τους ασκούμενους, για τους μαθητευόμενους, τίποτα όμως για τους δάσκαλους. Και την άλλη φορά θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα πρόγραμμα δασκάλων. Πρέπει. Δεν είναι αυτό μια κατηγορία προς τους δάσκαλους, αλλά είναι αναγνώριση πραγματικότητας. Λοιπόν, τελειώνω τώρα τη συζήτηση για τα δύο πρώτα θέματα. Θα περάσουμε τώρα στην καθηγήτρια κυρία Βίρεμαν. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους καθηγητές που μίλησαν πριν από μένα. Η, η, η, η Πρόεδρος ε, εκτός μικροφώνου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας μιλήσω σήμερα εδώ. Από τη σκοπιά της UNESCO μάλιστα, ιδιότερα της Γερμανικής Επιτροπής UNESCO. Και θα ήθελα καταρχήν να σας καταδείξω ποια είναι τα πολιτικά μέσα που έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η UNESCO για το σημερινό θέμα. Ποια είναι τα σημεία αναφοράς στα οποία μπορούν να αναφέρουν, να αναφερθούν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η UNESCO. Η Σύμβαση UNESCO για την πολιτισμική ε, πολυμορφία είναι κάτι που έχει δεχθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχει εντάξει στο δικό της νομοθετικό σύστημα και εξετάζουμε εδώ τα αποτελέσματα της Διεθνούς Διάσκεψης για την Κοινωνία της Πληροφόρησης και έθεσε τη σημασία της πολιτισμικής πολυμορφίας για την πολυμορφική κοινωνία. αυτή η πολιτιστική πολυμορφία, ταυτότητα, γλωσσική πολυμορφία και τοπικές ανάγκες είναι ένα μέσο που έχει προωθήσει η UNESCO. και αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η UNESCO εξετάζουν ε, τα, θέμα, τα θέματα αυτά όχι σαν κάτι κοινότυπο παραδοσιακό, αλλά πραγματικά σαν ένα τμήμα της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Είναι σημαντικά για την κοινωνία της γνώσης και το σύστημα αξιών στο οποίο ζούμε. Και γι' αυτό θα πρέπει οι πολιτικές ε, που στις οποίες βασίζονται όλα αυτά να είναι αντικείμενο έντονης μελέτης. Γενικά η UNESCO προωθεί ιδιαίτερα την ε, ανοιχτή πρόσβαση στις γνώσεις σε πολιτιστικά πολύμορφα περιεχόμενα κάθε είδους ανά τον κόσμο και αυτό βέβαια είναι και κάτι που ενδιαφέρει σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά που δεν είναι το αντικείμενο μας σήμερα. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε τρία θέματα. Καταρχήν, να σας πω δύο λόγια για τους στόχους που θα πρέπει να ακολουθεί μια πολιτική, κατά την άποψη της UNESCO, που επιτρέπει γενική προσέγγιση στο πολιτιστικό περιεχόμενο. Καταρχήν, είμαστε πεπισμένοι ότι η πρόσβαση σε μια πολιτισμική πολύμορφη κοινωνία είναι κάτι που ενδιαφέρει όλες τις κοινωνίες μας αλλά και που αφορά και τη δυνατότητα προώθησης ειρήνης και κοινωνικής συνοχής μεταξύ των κρατών μας. Ιδίως αυτές τις κοινωνίες που ζούμε σήμερα, στις ε, πολυπολιτισμικές δηλαδή. Ταυτόχρονα, βλέπουμε ότι μπορεί να προωθήσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση η ανταλλαγή αυτή των πολιτισμικών ε, περιεχομένων. Ταυτόχρονα όμως ο καθένας μας εμπλουτίζει τη ζωή του πάρα πολύ. Εάν μπορεί να γνωρίσει και να χρησιμοποιήσει για τον εαυτό του τους πολιτιστικούς ε, θησαυρούς άλλων λαών. Και τέλος, με την παγκοσμιοποίηση και τις προκλήσεις για τις θέσεις του μέλλοντος, είναι πιο, πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν εάν ξέρουμε και αναγνωρίζουμε την πολιτισμική κληρονομιά των χωρών μας. Και τέλος θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια πολιτική που προωθεί την πολιτισμική πολυμορφία και την ανταλλαγή θα πρέπει να είναι προς και εκείνων που δημιουργούν το περιεχόμενο αυτό το πολιτισμικό. Όχι μόνο στις μεγάλες γλώσσες, αλλά και σε μικρότερους ε, γλωσσικούς χώρους με πάρα πολλούς ενδυνάμει χρήστες μέσω του διαδικτύου. Αυτό έχει βέβαια επιπτώσεις και όσον αφορά την οικονομική ε, πρόοδο σε αυτές τις κοινωνίες. Τώρα ορισμένε παρατηρήσει όσον αφορά του κινδύνους που διαφαίνονται στο διαδίκτυο με τις πολιτικές αυτές που έχουν σαν στόχο πολιτισμικής ε, πρόθεσης και που απαιτούν οπωσδήποτε μεγάλες προκλήσεις. Καταρχήν θα μπορούσαμε να πούμε ότι στα τελευταία έτη είχαμε μια έντονη συγκέντρωση ισχύω στα χέρια λίγων μόνο διεθνών ε, επιχειρήσεων ΜΜΕ που πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τη συμπεριφορά τους. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, όπως τους λέμε gatekeepers, τυρορούς δηλαδή, που αποφασίζουν για την πρόσβαση στις υποδομές στο διαδίκτυο. Και έτσι δημιουργούν κατά κάποιο τρόπο διόδια όπου ο καθένας που θέλει να ωφεληθεί αναγκάζεται να καταβάλει τον οβολό του. Και παραδείγματος χάρη έχω κατά νου εδώ, όπως το Apple που ξεκίνησε με τα iTunes, με τη μουσική δηλαδή, και μετά ε, συσχετιζόμενο με το iPod και τώρα το iPhone. όπου όποιος θέλει να χρησιμοποιήσει όλα αυτά πρέπει να συμμορφωθεί με τους όρους της εν λόγω επιχείρησης, πράγμα που δεν είναι μόνο θέμα ε, οικονομικό, αλλά που σχετίζεται και με τα πρότυπα του περιεχομένου. Και αυτό σχετίζεται πια και με το θέμα της ελευθερίας σκέψεως και της ελευθερίας του τύπου. Oft, dass es eine ganze Reihe von Studien gibt zu einem Phänomen, UNESCO λοιπόν, απασχολείται και με ένα θέμα ότι η μεγάλη πολυμορφία που έχουμε στο διαδίκτυο δεν την χάνει εκμετάλλευσης. Ε, η UNESCO το αποκαλεί αυτό ε, ψευδή πολυμορφία γιατί δεν χρησιμοποιείται πραγματικά όλο το δυναμικό της πολιτιστικής πολυμορφίας. Και μόνο εκείνοι που πραγματικά ενδιαφέρονται επικοινωνούν και λίγο πολύ επιβεβαιώνουν τις απόψεις αλλήλων. Έτσι χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να αποχωριστεί κανένας από εκείνους που σκέφτονται διαφορετικά. Αυτή η αυτοαναφορά ορισμένων ομάδων στο διαδίκτυο θα πρέπει να εξεταστεί. Γιατί ίσως τελικά υποσκάπτει το ρόλο των οικογενειών και των σχολείων στην ε, μεταβίβαση της ιδέας της πολιτισμικής ταυτότητας. Αυτή τουλάχιστον είναι μια από τις ενισχύσεις της UNESCO. Και τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια ανησυχία ότι μπορεί αυτό το διαδίκτυο, τουλάχιστον νέα γενιά του διαδικτύου, να ε, οδηγήσει σε μια μεγάλη αγορά, όπου δηλαδή δεν θα έχουμε πολιτισμικά υψηλού επίπεδου περιεχόμενο προσβατό σε όλους, αλλά θα υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές για ψυχαγωγία στο διαδίκτυο τελικά ποιο θα είναι το μέλλον των, ε, του περιεχομένου υψηλού πολιτισμικού περιεχομένου και υψηλής πολιτισμικής αξίας ε, θα έχουν ευρεία πρόσβαση. Εδώ είναι ανησυχητικό αυτό, θεωρώ. Και σχετίζεται αυτό και με μια ε, συζήτηση για την ευρύτερη διεύρυνση των ε, δικαιωμάτων, πνευματικών δικαιωμάτων. Και αυτό μέσα στα πλαίσια μιας δίκαιης εξορρόπησης μεταξύ των ε, συμφερόντων των εκείνων που έχουν την πνευματική ιδιοκτησία και των χρηστών. Τι κάνει τώρα η UNESCO να υποστηρίξει όλα αυτά που σας παρουσίασα. Υπάρχει καταρχήν ε, αυτό το πρόγραμμα της UNESCO που λέγεται Information for All. Ενημέρωση για όλους. Ε, υπάρχουν εκεί ψηφιακές ε, <clears throat> βιβλιοθήκες που είναι ανοιχτές σε όλους χωρίς κόστος και γι' αυτό υποστηρίζει η UNESCO το Europeana σαν ένα παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής. Η UNESCO έχει ένα παρόμοιο πρόγραμμα, δηλαδή το World Digital Library που συμπληρώνει αν θέλετε το Europeana. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε πάντα τα δικαιώματα βηματικής τι γίνεται με τα έργα που δεν έχουν δημιουργό, τι γίνεται με την πολιτική της ανοιχτής πρόσβασης, open access, Σας έφερα και ένα εγχειρίδιο της γερμανική Επιτροπής UNESCO που έχει μεταφραστεί στα αγγλικά με ενίσχυση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δείτε τι εννοώ. Τελειώνω. Θέλω μόνο να αναφέρω το θέμα του πλουραλισμού των ΜΜΕ. Ήταν ένα σημαντικό τομέα της πολιτικής. Και ταυτόχρονα θα ήθελα να πω ότι η ΝΕΣΟ ενδιαφέρεται ιδιαίτερα οι κρατικοί, οι κρατικοί οργανισμοί ΜΜΕ να είναι διαθέσιμοι και στο διαδίκτυο σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βίντεμαν. Ο καθηγητής κύριος Ζων Ζωέλ Ζωνανή έχει το λόγο. Ελπίζω εσείς να είσαστε καθηγητής, να μην σας είπαμε καθηγητή χωρίς να είσαστε. Δεν έκανα λάθος. Είστε καθηγητής, μάλιστα. Το Google θα φταίει για την προφορά του ονόματος μου. Τέλος πάντων, κύρια Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ. Με μεγάλη ευγνωμοσύνη δέχτηκα να μιλήσω ενώπιόν σας σήμερα. Διότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ίντερνετ το θαυμαστό αυτό δώρο της τεχνολογίας πρέπει να αναρωτηθούμε αν είναι υπέρ ή κατά του πολιτισμού και δεν υπάρχει καλύτερο βήμα από το Ευρωπαϊκό Κενοβούλιο για να το αναρωτηθούμε αυτό. Αυτά που είπε η κυρία Βίλντεμαν ήταν ουσιώδη και ζωτικά. Είναι λογικές οι ανησυχίες αυτές μήπως ανεξέλεγκτα χωρίς καμία προσοχή από τις αρχές καταλήξουν όλα αυτά σε κάτι το αρνητικό. Θα αρχίσω υπενθυμίζοντας τρία νέα στοιχεία του θέματός μας και μετά θα καταρρύψω τρεις ψευδεστήσεις και τέλος θα αναφέρω τα τρία πράγματα που πρέπει να κάνουν οι αρχές για να ασκήσουν την ευθύνη τους. Θα μπορούσα να το κάνω ως ιστορικός διότι έτσι με, γι' αυτό με καλέσατε. καθώς ήμουν και διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας για πέντε χρόνια, είδα και εγώ ότι αυτή η Ευρωπαίανα βασίστηκε σε ελληνορωμαϊκές ρίζες. Θα συμπεθυμίζω ότι το θέμα μας είναι η σχέση του κοινού με τους δημιουργούς και τις δημιουργές. Καταρχήν, έχει υπάρξει μια εξέλιξη στις σχέσεις του κοινού με την χρονική πρόσβαση στα έργα, δηλαδή μια επιτάχυνση των τεχνολογιών που διακινεί τα πολιτιστικά έργα ταχύτερα και ακόμη περισσότερο, ακόμη ουσιοδέστερο υπάρχει το θέμα της ελευθέρωσης της πρόσβασης στα έργα ενώ παράλληλα <clears throat> η αποθήκευσή τους γίνεται όλο και πτητικότερη. Στο ραδιόφωνο ας πούμε. Η πρόσβαση του κοινού σε αυτό πώς γίνεται περίπου όπως αποθηκεύουμε βιβλία σε βιβλιοθήκες. Αλλά ο Μαλρό είχε πρώτος αναφέρει την ιδέα του φανταστικού μουσείου, αλλά τώρα κοντεύει να γίνει πραγματικότητα. Θα επανέλθω, θα επανέλθω. Και τέλος υπάρχουν διαφορετικές σχέσεις με, το, με τα έργα ολοκληρωμένα. Το ίδιο γίνεται και για τη μουσική. Δεν είναι σαν να βάζουμε απλώς μουστάκια στην τζοκόντα, γιατί αυτό είναι σπάνιο πια. Αλλά υπάρχει πια η δυνατότητα να δημιουργήσουμε νέα έργα μέσω της δημιουργίας αναμίξεων με παλαιότερα. Αποσπάσματα βέβαια. Όλα αυτά είναι καταπληκτικά αλλά μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσουν και σε αποβλάκωση. Γι' αυτό υπάρχουν οι τρεις ψευδεστήσεις που θα αναφέρω και που πρέπει να διαλύσουμε αν θέλουμε η, ο αυτός χαρακτήρας του καινούργιου αυτού εργαλείου να λειτουργήσει θετικά για τον πολιτισμό. Εννοώ για πεφωτισμένες δημοκρατίες βέβαια. Πρώτη ψευδέστηση η αποτελεσματικό και αφού μιλάω για τον πολιτισμό και την πολιτιστική αποτελεσματικότητα εννοώ για την πολιτική. Δηλαδή κατά πόσον είναι χρήσιμο ή όχι το αόρατο χέρι που έλεγε ο Αδάμ Σμιθ. Γιατί υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία και αύξηση των εγωιστικών συμφερόντων. Η εμπειρία της ιστορίας εδώ μας δείχνει ότι πράγματι συμβαίνει κάτι τέτοιο και ότι πρέπει να διαλύσουμε την ψευδέστηση αυτή. Η δεύτερη ψευδέστηση ότι η συλλογική δημιουργία είναι πια ο κανόνας και όχι η προσωπική. Βέβαια υπάρχουν όλο και περισσότερες ομαδικές εργασίες όπως τον κινηματογράφο και την τηλεόραση αλλά Νομίζω ότι πρέπει να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει και η προσωπική δημιουργία που καταλήγει στα καλύτερα και πολυτιμότερα έργα. Δεν είναι εδώ νομίζω ο καταλληλότερος χώρος και χρόνος για να αναφερθώ στο κατά πόσον στο διαδίκτυο τα συλλογικά έργα που διαδίδονται είναι από τα καλύτερα, δεν είναι το θέμα μας. Τρίτη ψευδέστηση και η χειρότερη από όλες. Ότι έχουμε τάχα μπει σε έναν κόσμο δωρεάν. Γιατί κάτι τέτοιο θα κατέληγε σε μία μείωση του πολιτισμού, θα κατέληγε σε ένα νεκροταφείο, πολιτιστικό νεκροταφείο. εξάλλου και στα μέσα του 19ου σε όλη την Ευρώπη μέχρι τη συνθήκη της Βέρνης είχε υποθεί ήδη ότι πρέπει τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών να προστατευθούν. Η δωρεάν παιδεία εδώ δεν υπάρχει. Πρέπει να αγοράζονται τα έργα Αυτό μπορεί να το κάνει κανείς ως φορολεγούμενος ή ως καταναλωτής και καταναλώτρια. Μη μου πείτε ότι αυτά που προσφέρει δωρεάν η διαφήμιση δεν τα πληρώνει ο φορολογούμενος και η φορολογούμενη. Το θέμα είναι ποια από αυτά τα κανάλια είναι το πιο αποτελεσματικό για να ευδοκιμήσει ο πολιτισμός. Και οι παρατηρήσεις αυτές με οδηγούν στα τρία συμπεράσματα. Στους τρεις πιθανούς ρόλους που μπορούν να παίξουν οι δημόσιες αρχές. Δηλαδή, πώς θα ασκήσουν καλύτερα τις ευθύνες τους δηλαδή. Οι δημόσιες αρχές με την ευρεία έννοια με την ευρία λεγόνια, οι δημοτικές αρχές, τέτοια πράγματα, πρέπει να συνδυάσουν την και το δημιουργία πλούτου και κέρδους με κάποια διευθέτηση όλων αυτών των αγορών. Δεν τα λέω από ακοβινική άποψη όλα αυτά. Γιατί ξέρω ότι ο πλούτος σήμερα δημιουργείται από δίκτυα, είναι δικτυακός πλούτος αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε ένα άλλο στοιχείο του χαρακτήρα της, τον, του ίδιου χαρακτήρα της φύσης των δημοσίων αρχών που είναι η παρέμβαση στο παιχνίδι. Και γιατί αυτό πρώτον, για να διασφαλιστεί η επιβίωση των έργων που διαδίδονται και στο διαδίκτυο και ψηφιακά διότι νομίζω ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στις επιχειρήσεις για να επιβιώσει η συλλογική μνήμη. Ένας ποιητής είχε πει «Ο κόσμος είναι γεμάτος φωνές που έχουν χάσει τα πρόσωπά τους». και συνεχώς τριγυρνάει ψάχνοντάς τα. Νομίζω ότι η αρχιοθέτηση των έργων στο δίκτυο, η ταξινόμησή τους είναι απαραίτητη για να μπορέσει κανείς να τα συμβουλευτεί και αυτό πρέπει να είναι ευθύνη των δημοσίων αρχών. Το λέω εδώ μέσα στο κοινοβούλιο όσο στεναρότερα μπορώ. Η αλλαγή των τρόπων αποθήκευσης πρέπει να εναπόκειται να διατύχει άνη διαχείριση από τις δημόσιες αρχές. Αλλιώς ποιος θα μας συγχωρήσει αν δεν έχουμε συντηρήσει, δεν έχουμε διατηρήσει όλα όσα δημιουργήσαμε. Πώς να ξέρουμε τι έγινε στις ευρωεκλογέ, ας πούμε αν δεν έχουμε περάσει από αποθήκευση των στοιχείων στη, στο διαδίκτυο. Αυτό ισχύει και για τη μουσική και για το ψηφιακό οπτικοακουστικό πεδίο όπως τα αρχεία που προτύπως δημιούργησε η Γαλλία για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Αυτά μπορούν να γίνουν με τη συμβολή των επιχειρήσεων αλλά χωρίς να έχουν εκείνες την αποκλειστική ευθύνη. Δεύτερον, τρία είπα θα αναφέρω δεύτερον. Δεύτερη ευθύνη των δημοσίων αρχών κατ' εμέ είναι να κατευθύνουν μέσα στο χάος και το χήμα τι γίνεται. Γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος που όλοι τον καταλαβαίνουν να μην μπορεί κανείς να βρει πια τίποτα. Το χήμα είναι ο κύριο απειλή της εποχής μας. Πρέπει να υπάρξει μια ιεράρχηση της προσφοράς. Δεν μπορούμε να δεχτούμε και αυτό να το κάνουν μόνο οι κερδοσκόποι και οι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις ή οι διαφημίσεις. Διότι έτσι ελκύεται μόνο η επιτυχία για την επιτυχία, ενώ ο πολιτισμός δεν βασίζεται στην επιτυχία αποκλειστικά. Αλλιώς θα έχουμε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον. Δηλαδή σε όποιον έχει θα δώσουμε παραπάνω, αλλά σε όποιον δεν έχει θα πάρουμε και ό,τι λίγο έχει. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια ιεράρχηση και η ιδιοφυής δημιουργοί του Google που κάπως τα άλλαξαν τα πράγματα από την ίδρυση μέχρι τώρα είχαν πει ότι αν αφήσουμε την διαφήμιση να ταξινομήσει την ε, προσφορά, τότε δεν θα έχει πια καμιά επιλογή ο καταναλωτής ούτε η καταναλώτρια. Ας πούμε για τα κινητά τηλέφωνα, θα είχαμε σε αυτή την περίπτωση πρώτον τις μεγάλες εταιρείες και όχι τα, τις καλύτερες συσκευές. Θα μπορούσε να γράψει και μια έκθεση το κοινοβούλιο ας πούμε για τους κινδύνους που εμπεριέχει η οδήγηση με κινητό τηλέφωνο. Τέλος το τρίτο. Όπως είχε πει και η κυρία Βίλντεμαν, υπάρχει η αναγκαιότητα να καταπολεμήσουμε οποιοδήποτε ιδιωτικό μονοπόλιο και ολιγοπόλιο. Πράγμα το οποίο ζητάει από καιρό η UNESCO και αυτό μου φαίνεται πολύ σημαντικό. Αλλά πρέπει να το δεχτούμε όλοι. Να υπάρξει ποικιλότης και των γλωσσών εσείς στο Κοινοβούλιο το αποδείξατε ότι δίνετε σημασία στις γλώσσες. Πρέπει να ξέρουμε ότι τα ιδιωτικά συμφέροντα δεν έχουν όρια. Και δεν το λέω ηθικά αυτά, το διαπιστώνω απλώς αντικειμενικά. Αυτή είναι η δυναμική της οικονομίας. Εξάλλου και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Το έχουν καταλάβει από καιρό, αφού αυτοί δημιούργησαν πρώτοι τους νόμους αντιτράστ στην αρχή του 19ου αιώνα και πρέπει να μην το ξεχάσουμε ποτέ αυτό. Και αυτό που ισχύει για τις Ηνωμένε Πολιτείες σίγουρα πρέπει να ισχύσει και παντού. Πολλά κράτη έχουν συνείδηση. Εγώ έκανα πολλή προσπάθεια να οργανώσω μια σταυροφαρία όχι κατά του Google του ίδιου αλλά για να μην είναι το Google το μονοπόλιο των βιβλιοθηκών και με μεγάλη έκπληξη είδα ότι πολλοί δέχτηκαν την έκκληση αυτή και στην Ιαπωνία και στην Κίνα. Είπανε «Α, γίνεται δηλαδή να αντισταθούμε σε αυτή την τάση, μόνο, τη μονοπωλιακή τάση». Και παρακαλώ να μην νομίσετε ότι τα λέω όλα αυτά από αλαζονία. Το βιβλιαράκι που είχα γράψει γι' αυτό μεταφράστηκε σε 15 ολόκληρες γλώσσες και σχολιάστηκε πλανητικά. Παρακαλώ λοιπόν την Ευρώπη να τα συνειδητοποιήσει όλα αυτά και εξάλλου η Ευρωπαία να το κάνει. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια διευθέτηση για να στηριχθούν όλοι οι δημιουργοί, οι εκδότες, οι βιβλιοπόλε. Σας υπενθυμίζω ότι το Google, αφού μιλάω για το Google, έχει κάνει ολόκληρη και κανονική ληστεία δημοσιεύοντας ψηφιακά χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών τους με διάφορα βιβλία. Αυτό είναι η φυσική αλαζονία των ιδιωτικών συμφερόντων. Ένα τέτοιο μονοπόλιο δεν θα ήταν ευκταίο. Παρακαλώ κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε να μιλήσω ομά. Όλοι αντιμετωπίζουμε εδώ αυτή την πρόκληση και πρέπει να προσέξουμε τρεις πειρασμούς να αποφύγουμε. Πρώτον, να θεωρήσουμε ότι η Ευρώπη είναι ξεπερασμένο πλαίσιο αντίδρασης προς την παγκοσμιοποίηση που διευρύνει με την πρόσβαση αλλά επίσης μειώνει τις ιδιαιτερότητες και αυτό θα μείωνε και τις ελευθερίες μας και τις διαφορές μας και την υποδειγματικότητα που θέλουμε να έχουμε και που έχουν η Κίνα, η Ιαπωνία και ο αραβικός κόσμος σε μας προβλέπει με τη δημιουργία της βιβλιοθήκης της Αλεξανδρίας ας πούμε. Άλλος πειρασμός που τον ξέρουμε πολύ καλά είναι η παρέτηση. Η παρέτηση έρχονται εδώ διάφοροι κύριοι και μας λένε δεν γίνεται τίποτα, ναι, πάει, πάει, δεν γίνεται τίποτα. Αυτή την παρέτηση αν τη δεχτούμε δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Τελειώνω κυρία μου, τελειώνω, σας παρακαλώ. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό ο δεύτερος πειρασμός να πρέπει να αποφευθεί και τρίτον, τρίτον και τελευταίο πρέπει να πω ότι Έχω βγάλει τις ρόδες για την προσγείωση κυρία μου. Λοιπόν, δεν πρέπει να αποθαρρυνθούμε μπροστά στο μέγεθος της πρόκλησης αυτής. Σας κατευχαριστώ κυρία μου που με ακούσατε με τόση υπομονή. Σα ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Τώρα δεν μας μένει και πολύ χρόνο για συζήτηση. Ένα, ένα λεπτό καθένας παρακαλώ. Η κυρία Καμαΐαβατ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ich bin ευγνώμων προς τον καθηγητή Ζενενή και την δόκτωρα Βίντεμαν για αυτά που μας είπε. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι έχουμε αφενός το διαδίκτυο που μπορεί να καταστεί προ στήσει προσιτή προς όλους την ε, πολιτιστική πολυμορφία που έχουμε. Από την άλλη μεριά είδαμε όμως ότι υπάρχει μια μεγάλη αγορά που δημιουργείται που ακριβώς περιορίζει την ελεύθερη ε, πρόσβαση. Αν κατάλαβα τη δόκτωρα Βίντεμαν σωστά, ε, η UNESCO θέλει μια πιο ευρία έννοια της ανοιχτής πρόσβασης ε, που πάλι ερχόμαστε βέβαια σε σύγκρουση με το δίκαιο των πνευματικών δικαιωμάτων. Μπορείτε να μας πείτε κάτι για αυτό το εδώ. Ευχαριστώ. Κύριος Βάτιμο. Εκτός μικροφώνου. Εγώ ήθελα απλώς να ρωτήσω τους ομιλητές που μας είπαν τα όσα ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι σαφές αυτή τη στιγμή πώς έχει το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Διότι εγώ ξέρω ότι υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με το θέμα των ανταλλαγών peer-to-peer, ο ένας που ανταλλάσσει μουσική με τον άλλον χωρίς να πληρώσει δικαιώματα του δημιουργού. Ε, και θα ήθελα να ξέρω αν είναι σαφής η κατάσταση, γιατί δεν ξέρω καλά πού βρισκόμαστε. Ξέρω ότι στο Κοινοβούλιο έχουμε δύο Σουηδούς εκπροσώπους ε, από το κόμμα των πειρατών που δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να συναντήσω. Θα ήθελα να τους γνωρίσω. Δεν ξέρω όμως αν κάποιος είναι μέλος εδώ της Επιτροπής μας. Και το θέμα είναι το εξής. Ξέρουμε που βρισκόμαστε. Διότι αφενός έχουμε το θέμα των δικαιωμάτων των δημιουργών ε, των πολιτιστικών αγαθών που θέλουμε να αλλάξουμε και από την άλλη υπάρχει το θέμα της δημόσιας πρόσβασης ε, για όλους. Και όλες. Και όλες. Μπορούμε να φανταστούμε λοιπόν μία δημόσια δράση η οποία να αποζημιώνει με κατάλληλο τρόπο τους δημιουργούς, τους μουσικούς, τους καλλιτέχνες εν γέννη και από εκεί και πέρα να είναι διαθέσιμα για όλους τα πολιτιστικά αγαθά. Παραδείγματο χάρη στο θέμα των δικαιωμάτων του δημιουργού υπάρχει κάποιο χρονικό όριο στο οποίο λήγουν τα δικαιώματα. Μετά από 50 χρόνια, για παράδειγμα, οι κληρονόμοι του Πυραντέλου και του Κάφκα δεν έχουν πνευματικά δικαιώματα, δεν χρειάζεται να λαμβάνουν κάτι. Ε, πώς μπορούμε να αντιδράσουμε. Αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημα. Κατά τα άλλα η τεχνολογία μας βοηθά, αλλά πρέπει ε, να ε, συμφιλιώσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Κύριος Μπόρις, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα που θίξατε. μετά από την ατμομηχανή και τις υπόλοιπες επαναστάσεις ε, ήρθε και η επανάσταση του διαδικτύου. Βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλές απειλές και προκλήσεις, ε, μπορεί να αποτελέσει και ένα ε, μέσο επικίνδυνο. Μπορεί να μεν αυτή τη στιγμή να είναι παγκόσμιο μέσο που ε, βοηθά την ε, ενημέρωση προς όλους, αλλά διαρωτώ με μήπως θα πρέπει να γίνει μια ανάπτυξη σαν τη δημόσια τηλεόραση, χωρίς σύνορα. Βέβαια το διαδίκτυο δεν έχει κανένα δίκτυο. Είναι ένα μέσο <clears throat> ελευθερίας και κοινοτομίας άλλοι τομεί εξελίσσονται έτσι γιατί δεν έχουν καθόλου σύνορα, δεν έχουν όρια, δεν υπάρχουν οι περιορισμοί που είχαμε στο παρελθόν και που περιορίζαν την εξέλιξη, σύνορα, όρια κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να έχουμε μια σωστή ισορροπία. Α, δηλαδή το μονοπόλιο να μην επικρατήσει πάνω στην αγορά του διαδικτύου. Η σύμβαση της ε, ε, ε, ε, καθορίζει και διέπει τα πνευματικά δικαιώματα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κανένα ιδανικό σύστημα ισορροπίας. <clears throat> Μια ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δικαιωμάτων του δημιουργού και της ελευθερίας των χρηστών του διαδικτύου. Παραδείγματος χάνει σε συστήματα όπως το music sharing και άλλα παρόμοια. Θα πρέπει νομίζω να έχουμε ένα σύστημα όπου να προστατεύονται τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπου οι δημιουργοί να μπορούν να πληρώνονται για την ε, απόδοσή τους, ταυτόχρονα όμως οι χρήστες του διαδικτύου να ξέρουν ότι δεν επιτρέπεται να καταπατούν αυτά τα πνευματικά δικαιώματα. Χρειαζόμαστε νομίζω να θέσουμε σε ισχύ ένα τέτοιο σύστημα που να είναι αποδεκτό για όλους. Βέβαια οι χρήστε του διαδικτύου θέλουν όλα να τα έχουν δωρεάν ε, στο διαδίκτυο. Αλλά αν δεν έχουμε ένα τέτοιο σύστημα, τότε δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θα πρέπει να κάνουμε και για του δημιουργού. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Τώρα εγκαταλείπουμε κάπως το θέμα της ε, ακροασής μας. Αυτά τα θέματα εξάρτητα στη βιομηχανία, η τρες, η νομική, λίγο και σε εμάς γιατί το σημερινό μας ε, θέμα είναι εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διαπολισμική κατανόηση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί και να μην περάσουμε σε όλα αυτά τα προβλήματα για το copyright, για τα πραγματικά δικαιώματα που έχουμε να συζητήσουμε στην θητεία μας. Θα ήθελα να παρακαλέσω τώρα να απαντήσουν ε, οι δύο ομιλητές, η κυρία Βέντεμαν πρώτα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω κάτι για την ελεύθερη πρόσβαση, το open access που ανέφερε η κυρία Βουλευτής. Αυτή η αρχή δεν είναι σε σύγκρουση με το ισχύον δίκαιο πνευματικών δικαιωμάτων, ε, γιατί ε, δικαιώματα που έχουν δημιουργηθεί μπορούν να καλυφθούν με χρήματα και να είναι τα έργα αυτά προσβατά. Αυτό δεν ε, διακυβεύει τα δικαιώματα των δημιουργών, αλλά είναι μια συγκεκριμένη πολιτική που ακολουθείται. Γιατί τι το θέμα κατά πόσον υπάρχει κάποιο περιεχόμενο το οποίο δεν επιτρέπεται να τύχει μιας εκμετάλλευσης δηλαδή να υπάρχει ένα σταθμός διοδίων όπως είπατε και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατόπιν ε, καταβολής ενός τέλους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάτι παρόμοιο υπάρχει στους ε, κρατικούς ε, οργανισμούς ΜΜΕ που υπάρχει ένα κόστος αλλά το κόστος καλύπτεται το κράτος. Τίποτα δεν είναι χωρίς κόστος. Δεν υπάρχει λοιπόν εδώ αντίφαση μεταξύ της ελεύθερης πρόσβασης και του ισχυόντος δικαίου για πνευματικά δικαιώματα. Ακριβώς, ε, παραδείγματος χάρη, ε, στο στο δομέα της κρατικής τηλεόρασης ο χρήστης πληρώνει κάθε μήνα ένα τέλος και το είπε και η UNESCO ότι και το διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό μέσο ενημέρωσης που ε, θα πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες αυτές τις πληροφορίες χωρίς συμπληρωματικό τέλος. Όλα αυτά είναι σημαντικά σε σχέση με το ότι εκτός από τα διάφορα ε, επιχειρησιακά μοντέλα που είναι δυνατά, δεν τα καταδικάζει κανένας, Θέλουμε να φροντίσουμε ορισμένα περιεχόμενα υψηλής πολιτιστικής αξίας που είναι σημαντικά και την παιδεία θα πρέπει να είναι ε, πρόσβατα σε όλους. Αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει και τη δική σας επιτροπή ιδιαίτερα. Δηλαδή πέρα από την ψηφιακή βιβλιοθήκη, πέρα από το σχέδιο της Ευρωπαϊκά, να δούμε ποια είναι η πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιεχόμενο στον δημόσιο τομέα που διατίθεται ελεύθερα και όχι μόνο στα πλαίσια της ψηφιακής ατζέντα όσον αφορά την εμπορική χρήση. Θα ήθελα να απάντησε και σε βάση κατά πόσον ε, υπάρχει σαφήνεια. Όλα είναι αυτή τη στιγμή εν ροή. Η προσπάθεια μου ήταν να διευκρινίσω ότι αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε υπάρχει μια τάση που έχει προβλεφθεί, που ενδυναμώνεται, που πραγματικά εμφανίζεται αυτή τη στιγμή έντονα λόγω της οικονομικής η ε, οικονομικής προσέγγισης των δικτύων αυτών ε, Economies of Scale and Scope όπως το λέμε αναφέρθηκε το Apple αλλά υπάρχουν και άλλα όπου δεν υπάρχει μόνο εκμετάλλευση μιας ε, ειδικής ηγετικής σχέσης, ε, σε θέσεις συγγνώμη, στην αγορά, αλλά και στις λεπτομέρειες μια επιχείρηση. Όπελ το κάνει αυτό. Εμείς επιτρέπουμε μόνο πρόσβαση πληροφοριών που ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένη γραμμή, αν θέλετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό σε σχέση και με την ελευθερία του τύπου. Αυτό είναι ένα νέο φαινόμενο και θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. και να σκεφτούμε λιγάκι τι θέλουμε για την Ευρώπη ακριβώς. Και εδώ θα ήθελα να αφαιρθώ και σε αυτό που είπε ο καθηγητής κ. Ζερανή. Ότι πραγματικά στην Ευρώπη έχουμε ένα ρόλο παραδειγματικό να παίξουμε. Υπάρχουν πάρες πολιτικές που παρουσιάζονται. Τώρα τι θα γίνει από εκεί και πέρα δεν ξέρω, δεν πρέπει να ξανεφεύρουμε τον τροχό. αλλά όπως καταλαβαίνουμε εμείς την πολιτιστική πολυμορφία και την πολιτιστική ανάπτυξη πολλά μπορούμε να κάνουμε νομίζω ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Όπως και εσείς κυρία μου, νομίζω ότι δεν χρειάζεται εδώ να αρχίσουμε μια ολόκληρη νομική συζήτηση για τα πνευματικά δικαιώματα. αλλά δεν μπορεί και να αποφύγει η Επιτροπή σας τουλάχιστον να θέσει τα πολιτικά και οικονομικά προβλήματα. Ως ιστορικός εντυπωσιάστηκα από τις συζητήσεις που έγιναν στα μέσα του 19ου αιώνα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Καταρχήν δύο σχολές μάλλον μέχρι να βρεθεί η ισορροπία που είπατε κύριε μου. Οι μεν έλεγαν δεν υπάρχει δημιουργία που να μην στηρίζεται σε προϋπάρχοντα υλικά. Άρα δεν μπορεί να υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα, όλα πρέπει να είναι δωρεάν. Οι που ήταν οι φιλελεύθεροι οικονομολόγοι έλεγαν ότι ο δημιουργός ενός έργου πρέπει αιωνίως να διατηρεί τα δικαιώματα και να τα έχουν και από απόγονοί του. Και τελικά βρέθηκε μια, ένας συμβιβασμός αυτής της πεντηκονταετίας των πνευματικών δικαιωμάτων Επίσης πρέπει να παρατηρήσουμε ότι μερικοί λέγανε τότε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων και ότι καλά ήταν ως ιδέα αλλά στην πράξη δεν γίνεται, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Και ότι και να υπήρχε νόμος δεν θα γινόταν σεβαστός. Μπορεί, αλλά μετά από μερικές γενναίες καταλήξαμε στη σύμβαση της Βέρνης Πού το κατάφερε αυτό. Και σήμερα όμως ισχύει ότι πρέπει ένας δημιουργός να μπορεί και να επιβιώσει από τα έργα του. Εκτός αν είναι ήδη πλούσιος. Άρα οι πτωχότεροι δεν θα δημιουργούν. Ή θα πρέπει να τον βοηθούν διάφοροι με κίνες και άρα θα έχουν και δικαίωμα λογοκρισίας. Πρέπει να το σκεφτούμε όλοι μας αυτό το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων την εποχή του ίντερνετ. Να μην απογοητευτούμε, να μην αποθαρρυνθούμε. Υπάρχουν δυνατότητες μικροπληρωμών και απ' την άλλη φυσικά πάντοτε θα υπάρχουν και οι υποκλοπές. Νομίζω ότι όπως και στα έργα Western με τον Γκάρι Κούπερ πρέπει τελικά να εμφανιστεί ο Σερίφης. Αυτό ισχύει και για τους δημιουργούς και για τους χρήστες και τις χρήστριες. Πρέπει όμως να υπάρξει ρόλος και για τους μεσολαβητές που να δώσουν τη δυνατότητα και μεσολαβήτρες που να δώσουν τη δυνατότητα στο κοινό να καταλάβει τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και εννοώ εδώ τους δασκάλους και τις διδασκάλισες. Νομίζω ότι ως πανεπιστημιακοί πρέπει και εσείς, αναφέρομαι στους προηγούμενους ομιλητές, να καταλάβετε τη σημασία των πνευματικών δικαιωμάτων και για να πω και ένα αστιάκι. Όταν ακούγαμε μαθήματα στο ραδιόφωνο, μαθαίναμε το ρητό μακάρια τα ποτάμια που μπορούν να ακολουθούν τον ρούν τους στα γαλλικά και τα μαθήματά τους από την κήτη τους δηλαδή, το κρεβάτι. Τέλεια. Ωραία. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Εκτελεστική Επιτροπή. Δύο λεπτά παρακαλώ μόνο. Ο κ. Σακέτη. Δύο μινούτι. Yes. Ε, thank you. Thank you for this. Ε, Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σήμερα το πρωί αναφέρθηκε ότι ελοχεύουν κίνδυνοι, ότι υπάρχουν απειλές και υπάρχουν και ευκαιρίες για τη χρήση της νέας τεχνολογίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η σωστή κίνηση για να ελοχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι και να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες είναι το να γνωρίζουμε το θέμα. Ε, σε αυτή την περίπτωση να γνωρίζουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λίγα πράγματα για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτή τον τομέα πολιτικής, ο οποίος νομίζω ότι είναι συμπληρωματικός ε, με τα θέματα τα οποία συζητήσαμε σήμερα. Η πρώτη πρόκληση πριν από 4-5 χρόνια όταν ε, αρχίσαμε να ασχολούμαστε με αυτό τον τομέα ήταν να έχουμε ένα κατάλληλο ορισμό με τη βοήθεια μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων καταλήξαμε σε έναν ορισμό για το media literacy και βασίζεται σε τρεις βασικούς στόχους και τρεις βασικές ικανότητες. Καταρχάς, η ικανότητα πρόσβασης και χρήσης του διαδικτύου. Δεύτερον, η σωστή αξιολόγηση του περιεχομένου που προσφέρουν τα μέσα. Και τρίτον, κάτι πολύ σημαντικό σήμερα, η δυνατότητα να επικοινωνούμε και να χρησιμοποιούμε τα ε, μέσα αυτά με δημιουργικό και ενεργό τρόπο. Φυσικά βέβαια θεωρούμε ότι το media literacy σχετίζεται με όλα τα μέσα ε, και τη τηλεόραση, το ραδιόφωνο, την ηχογραφημένη μουσική, τα έντυπα μέσα, το διαδίκτυο και άλλες ε, τεχνολογίες ψηφιακής μετάδοσης. Θεωρούμε ότι πλέον το media literacy αποτελεί πολύ σημαντικό παράδειγμα για να είναι κάποιος ενεργός πολίτης. Αλλά διαδραματίζει και ουσιαστικό ρόλο στο, στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και στην ταυτότητά μας. Αυτοί που γνωρίζουν καλά τα μέσα μπορούν να κάνουν πιο ενημερωμένες επιλογές. και ως προς την αγορά πολιτιστικού περιεχομένου. Επομένως, οι πολίτες που έχουν πολύ μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας γιατί έχουν τα μέσα να επιλέξουν τι θα δουν και τι θα διαβάσουν ε, θα γνωρίζουν πολύ καλύτερα και τις συνέπειες των επιλογών τους και νομίζουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Η κυρία ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας ε, για αυτή τη δημόσια κρόαση. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη, η οποία υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Μαΐου του 2010 και αυτή η ψηφιακή ατζέντα περιλαμβάνει μία σειρά από δράσεις ε, και ο τελικός στόχος είναι να βγει η Ευρώπη από την κρίση. Μεταξύ των δράσεων, ε, οι οποίες είναι κατανεμημένες σε 7 τομείς, περιλαμβάνονται και αυτά που μόλις ανέφερε ο συνάδελφος, και πιο συγκεκριμένα θέλουμε να θεμελιώσουμε το να γνωρίζει κάποιος και να μπορεί να διαχειριστεί ε, την ψηφιακή τεχνολογία. Δηλαδή θέλουμε να συμπεριλάβουμε την ηλεκτρονική μάθηση στις ε, εθνικές πολιτικές ε, παιδείας. Κάποια άλλα στοιχεία που καθορίζονται σε αυτή την ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη είναι να έχουμε τα μέγιστα δυνατά ωφέλη για την κοινωνία από την εφαρμογή της ε, τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας και αυτό συμπεριλαμβάνει και την ανάπτυξη της Ευρωπαίαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου έχει το λόγο. Ο κ. 10. Please, two minutes. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, καθηγητές, διδάκτορες εδώ. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ εξ ονόματος της Ισπανικής Προεδρίας. Πρέπει να πω ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν συνειδητοποιήσει πλήρως τα θέματα που συζητάμε σήμερα εδώ στην Επιτροπή σας. Εσείς προσπάτως εδώ εγκρίνατε ένα ψήφισμα για την ε, ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο διαδίκτυο που επισημαίνεται πόσο σημαντικά είναι τα θέματα αυτά. Από πλευρά Συμβουλίου πρέπει να σας πω ότι η ανησυχία για τα θέματα αυτά υλοποιείται σε αυτά παραδείγματα. Να σας υπενθυμίσω ότι η Τσεχική Προεδρία πέρσι, το Μάιο του 2009, ενέκρινε ένα έγγραφο για την εκπόνηση ενός στρατηγικού πλαισίου για την ψηφιακή τεχνολογία για το 2020 και εκεί καθορίζονται καταρχάς ε, οι δυνατότητες ε, της ε, ενδυνάμωσης της, επί, της παιδείας και επίσης η ανταγωνιστικότητα και η δημιουργικότητα. Επίσης αναφερόμαστε και στις γλωσσικές προκλήσεις για τους μαθητές, καθώς επίσης και την πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα στο διαδίκτυο. Σε αυτό το στρατηγικό πλαίσιο λοιπόν για την ε, παιδεία και την ενημέρωση, η Ισπανική Προεδρία είχε την τιμή να ετοιμάσει στη διάρκεια των εργασιών της κάποια συμπεράσματα, τα οποία ναι μεν αναφέρονται επιγραμματικά, αλλά λαμβάνουν υπόψη τα θέματα αυτά. Ε, στις 26 Μαΐου ε, δημοσιεύτηκαν αυτά τα συμπεράσματα και εκεί αναφέρεται και η κοινωνική διάσταση της παιδείας αλλά και η διεθνοποίηση ε, των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά ταυτόχρονα και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης ε, η οποία πλέον είναι συνειφασμένη με τις γλωσσικές δεξιότητες και τις δυνατότητες πρόσβασης στην ε, τεχνολογία και την πληροφορική. Θα πρέπει επίσης ε, να πω ότι όταν ήρθε εδώ ο Υπουργό ε, Παιδείας, ο οποίος στάθηκε σήμερα το απόγευμα, είχε ήδη επισημάνει πόσο σημαντικό θεωρεί το θέμα αυτό η Ισπανική Προεδρία και τα θέματα δηλαδή που σχετίζονται με τις ψηφιακέ δεξιότητες των μαθητών και των φοιτητών, αλλά και τα γλωσσικά θέματα. Ένα τελευταίο αίτημα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Βελγική Προεδρία, η οποία θα αναλάβει τα ενία σε λίγο, θα έχει ένα θέμα το οποίο θα είναι αφιερωμένο στα σχολεία του 21ου αιώνα και αναφέρεται και στις ε, ψηφιακές δεξιότητες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Καρσάζα από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ισπανίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θα ήθελα απλώς να συμπληρώσω ε, τα όσα ακούσαμε σήμερα εδώ και να αναφερθώ στις πτυχές ε, που επεξεργαστήκαμε και εμείς ε, στο Συμβούλιο και σχετίζονται με τον πολιτισμό και με τα οπτικοακουστικά θέματα. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει απόλυτο συντονισμό στο Συμβούλιο με τα όσα συζητήθηκαν εδώ σήμερα και με τι εργασίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μία από τι μεγαλύτερε προκλήσει, γιατί θεωρώ ότι αυτέ είναι κοινέ προκλήσεις, ε, ήταν να προχωρήσουμε ένα από τα προγράμματα που θεωρούμε ότι είναι υψή τη σημασία και που ε, ακολουθήσαμε από τα πρώτα του βήματα, όπω είπε και ένα από του προλαλήσαντε πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε και να τελειώσουμε το πρόγραμμα της Ευρωπαϊάνα εγκρίθηκαν τα συμπεράσματα στις 10 Μαΐου, τα οποία συμπεράσματα τονίζουν ότι το να ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα σημαίνει ότι ε, θα πρέπει να καθορίσουμε και τι Ευρωπαία θέλουμε να έχουμε και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει αυτό το πρόγραμμα. Μία από τις βασικές πτυχές που θεωρούμε ότι είναι σημαντικές είναι να αυξηθεί το ψηφιακό περιεχόμενο, μία δέσμευση που πρέπει να θεωρήσουν προτεραιότητα όλα τα κράτη-μέλη στις πολιτικές τους, αλλά επίσης θα πρέπει να συμπληρώνεται και με τη συμμετοχή των ε, ε, πολιτιστικών φορέων, που είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν ζωή στο πρόγραμμα της ναι. Ευρωπαϊκής. Επίσης η έμφαση στο χρήστη, ε, που νομίζω ότι είναι αλληλένδετο με αυτό που ακούσαμε εδώ σήμερα το διαδίκτυο επιτρέπει αυτές τις ανταλλαγές, ε, την επικοινωνία και τη ζωντανή εξέλιξη του περιεχομένου και δεν μπορούμε να χαθούμε, ε, ε, να χάσουμε αυτό το σημείο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής. Θα πρέπει επίσης να εξοικειωθούν οι χρήστες και να αυξηθεί η γνώση που έχουν επί του θέματος και να το διασυνδέσουμε με έναν από τους βασικούς στόχους που αναφέρθηκαν εδώ σήμερα, η παιδεία. Ο πολιτισμός ως ε, αναπόσπαστο κομμάτι της παιδείας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα τώρα να κλείσουμε εδώ την ακρόαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες που ήρθαν εδώ για τον κόπο τους να έρθουν εδώ, να μας παρουσιάσουν τις απόψεις τους και έστω και τόσο σύντομα όλοι δημιουργήσαμε κάποια εντύπωση όσον αφορά τις δεσμές που υπάρχουν. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι έχετε μπροστά σας ανθρώπους που θέλουν να εκμεταλλευτούν τις γνώσεις σας και που θέλουν στο υπόλοιπο της ε, νομοθετικής θητείας να δράσουν στον τομέα αυτού, αυτό όπου μπορεί να το κάνει το ευρωπαϊκό επίπεδο. Και Είχαμε λόγο να έχουμε το Συμβούλιο εδώ, γιατί πολλές σοφές αποφάσεις λαμβάνονται στο Συμβούλιο. Η εφαρμογή τους όμως καμιά φορά υστερεί ή και λείπει. Και γι' αυτό ε, χαίρομαι που ε, το Συμβούλιο είπε από μόνο ότι θα πρέπει να εφαρμόζει ε, στις πατρίδες, ε, στα κράτη-μέλη, αυτά που εμείς εδώ αποφασίζουμε. Αυτό είναι σημαντικό για μας, όλους τους πολίτες, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Σας ευχαριστώ. Ε, μια που είμαι μόνη μου εδώ, δεν μπορώ καν να σας σφίξω το χέρι. Ε, ελπίζω να δείξετε κατανόηση, σας εύχομαι καλή επάνωδο και εμείς συνεχίζουμε. Σημείο 7 της ημερησία διάταξη. Κρατικά θεραπευτικά μέσα στην πληθυακή εποχή. Το μέλλον του διτού συστήματο. Εισηγητή είναι ο Ιβο Μπέλετ. Το έχει παρουσιάσει πολύ συχνά το θέμα. Έχει το λόγο, Ιβο. Hartelijk dank, Doris. Ik zal een, mijn, mijn inleiding zo kort als mogelijk houden en zo concreet mogelijk om nog zoveel mogelijk ruimte voor de discussie te laten hier op het late middaguur. Eerst en vooral dus... Θα ήθελα να σας αναφέρω την κατάσταση της εξέτασης της έκθεσής μου όσο δυνατόν συντομότερα. Καταρχήν, το θέμα έχει πολλές πτυχές που δεν θα τις αναφέρω όλες στο έγγραφο εργασίας γιατί διότι πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας ιδιαίτερα στο θέμα στο εύρος της εντολής που μας έχει δοθεί παραδείγματος χάρη δεν θα μιλήσω για τα blog για την νομική ευθύνη που μπορεί να υπάρχει για ορισμένες δραστηριότητες όπως liability to reason περιοριζόμαστε δηλαδή στο θέμα ακριβώς που αναφέρει η έκθεση μου. Είχαμε πολλές αντιδράσεις από ενδιαφερόμενους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, προσώπους του τύπου, και τις προσέξαμε όλος ιδιαιτέρως. Το έγγραφό μας λοιπόν τροποποιήθηκε αναλόγως και θα συνεχίσουμε να το χτενίζουμε. με βάση ό,τι πληροφορίες μας δοθούν. Δεύτερον, εδώ χρειάζεται κάποια εξισορρόπηση γιατί ορισμένες χώρες μέλη των οποίων λειτουργεί λίγο πολύ καλά ο δημόσιος τομέας Οφελείτε, ε, ωφελούνται από την περασμένη ανακοίνωση της Επιτροπής αλλά δεν ισχύει το ίδιο και για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπου Ακούγονται πολλές επικρίσεις για τα δημόσια δίκτυα αναμετάδοση, ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία, αλλά και ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα χρεοκοπίας τους. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να τα συνδυάσουμε αυτά. Δύσκολο πράγμα. Όσοι εισηγητής δεν θέλησα να εφαρμόσω την μέθοδο naming and shaming γιατί έτσι δεν θα είχαμε αξιόπιστα αποτελέσματα. Αλλά επειδή δεν επιλέξαμε αυτή τη μέθοδο, επιλέξαμε μια δομική ανάλυση γνωρίζοντας πολύ καλά ότι το θέμα δεν είναι να καταλήξουμε σε μία ομοιόμορφη λύση για όλους, αλλά σε μία διαφοροποιημένη πρόταση. Τρίτον, πολύ σημαντικό, οι σχέσεις καταρχήν της τηλεοπτικής και ψηφιακής γενικότερα αναμετάδοσης με τον γραπτό τύπο Για μερικούς υπάρχει θέμα του ανταγωνισμού, για άλλους όχι. Άλλοι δηλαδή είναι πολύ ικανοποιημένοι από τη διάδοση ηλεκτρονικός των μέσων και του γραπτού τύπου. Πώς μπορούμε λοιπόν να αντιδράσουμε και να βοηθήσουμε Οι συνάδελφοι μου έκαναν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και θα τις αναφέρω εδώ. Ορισμένες μόνο. Λοιπόν, το σημείο 9 υπήρξε πολύ αμφιλεγόμενο γιατί εκεί γίνεται λόγος για το Ευρωπαϊκό Παρατήριο των Οπτικοακουστικών από το οποίο ζητούμε να ελέγχει αν τα κράτη-μέλη σέβονται τα πρότυπα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί ενδιαφερόμενοι, το παρατήριο αυτό βεβαίως δεν θα ελέγχει, θα παρατηρεί απλώς. Γιατί ο έλεγχος είναι δουλειά των κρατών μελών, αυτό δεν το αμφισβητούμε. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν είναι το παρατηρητήριο αυτό που εδρεύει εν Στρασβούργο να επαληθεύει για τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που είναι όλα και μέλη της Ένωσης και συνυπέγραψαν τη σχετική δήλωση, να τους ζητήσει λοιπόν να παρατηρούν σε ποιο βαθμό τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης σέβονται τις ίδιες τους τις συστάσεις. την ανεξαρτησία των σταθμών και τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότησή τους διότι εάν ο προϋπολογισμός μερικών σταθμών εγκρίνεται από το κοινοβούλιο τότε δεν είναι ανεξάρτητο ο σταθμός. Και τέτοια πράγματα πρέπει να επαληθεύει το παρατηρητήριο. Και για να τελειώσω τώρα, στην παράγραφο 12 γίνεται λόγος για διαφάνεια ως προς την ιδιοκτησία των σταθμών εκπομπής. Και εδώ ακούσαμε πολλές αντιδράσεις. Λογικό αυτό. Ιδίως για τους ιδιωτικούς σταθμούς. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχε, πει, είχε δηλώσει ότι πρέπει στο ψήφισμά μας ότι στο ψήφισμά μας δεν είχαμε αξιόπιστα στοιχεία. Τους απαντώ όμως ότι η Κομισιόν χρησιμοποίησε μια μελέτη και εκείνη από το 2008 που και εμείς δεν ξέρουμε πόσο αξιόπιστη είναι γιατί δεν την έχουμε δει και θα θέλαμε να τη συζητήσουμε όπως το είχε εξάλλου αναγγείλει να μας προτείνει ένα πλήρες σχέδιο δράσης με βάση τους δείκτες που θα, έχει, που θα έχουν προκύψει από τη μελέτη για να καταλάβουμε και εμείς καλύτερα ποιες είναι οι ιδιοκτησιακές δομές των ιδιωτικών σταθμών αναμετάδοσης. Θα μπορούσα να πω και άλλα, αλλά δεν θα τα πω για να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφος Κύρκοπ. Uh, thank you very Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέλετ. Έκανε πολύ σκληρή δουλειά για αυτή την έκθεση και πολλά από αυτά που έχει συμπεριλάβει είναι πολύ θετικά. Η έκθεση αυτή εστιάζει κυρίως ε, στις δημόσιες μεταδόσεις, αλλά αν δούμε και τα ε, άλλα συστήματα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν ε, και στενές σχέσεις μεταξύ δημοσίων και εμπορικών μεταδόσεων και να αναγνωρίσουμε και τις δυσκολίες της δεύτερης κατηγορίας. Να αναφερθώ καταρχάς σε ένα συνδυασμό του σημείου 11 και της αιτιολογικής σκέψης K, όπου αναφέρεται τα προβλήματα τα οποία απειλούν ε, ε, τη ζωή των δημόσιων μεταδόσεων που είναι και πολιτικά και οικονομικά. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια οικονομική κατάσταση και ε, αυτή τη στιγμή που δημιουργεί τα ίδια προβλήματα και για τις δημόσιες υπηρεσίες ενημέρωσης και για τις ε, ιδιωτικές. Επομένως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις επιπτώσεις που υπάρχουν ε, για τις ε, δημόσιες υπηρεσίες ενημέρωσης. Αναφέρεται επίσης ότι ο κατακαιρματισμός του κοινού είναι από μόνος του κόσ. Εγώ δεν συμφωνώ. Ο κατακαιρματισμός είναι ένας όρος, αλλά το άλλο θέμα είναι ότι είναι θέμα επιλογής. Εάν κάποιο, αν θέλει να δει τηλεόραση, ε, μπορούμε να πάρουμε το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ναι, μεν η ψηφιακή και δορυφορική τηλεόραση ε, άρχισε με πολύ αργό τρόπο. Τώρα όμω άρχισαν να έχουμε καινοτομίε και στι αθλητικέ μεταδόσει και στη ψυχαγωγία εν γέννη. Και αυτή τη στιγμή τα δημόσια μέσα ενημέρωσης ε, προσπαθούν να αλλάξουν το πρόγραμμά τους γιατί βλέπουν ότι μοιράζονται ε, το μερίδιο της τηλεθέασης με την ιδιωτική τηλεόραση και θέλουν περισσότερους θεατές. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ ευαίσθητη ισορροπία οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τελικά πάντα επιλογή του παρόχου. Εδώ, για παράδειγμα, στις Βρυξέλλες, ακόμα στους Δήμους, οι ε, πάροχοι τηλεοπτικών δικτύων δεν μπορούν να έχουν ανταγωνιστικό ρόλο. Σας υποχρεώνουν να επιλέξετε τον ένα και μόνο πάροχο που παρέχει τηλεόραση στο Δήμο. Και αυτό φυσικά ε, είναι ε, κατά των συμφερόντων των ίδιων των επιχειρήσεων. Φαντάζομαι ότι όλοι μας εδώ στη ζωή μας έχουμε πρόσβαση σε εκατοντάδες ε, τηλεοπτικά κανάλια. Ίσως είμαι παραδοσιακός εγώ, αλλά θεωρώ ότι το μεγαλύτερο τμήμα του περιεχομένου αυτών των καναλιών που βλέπουμε είναι άχρηστο. Δεν θεωρώ βέβαια ότι αυτό είναι επαρκής αιτιολόγηση να περιορίσουμε το προσφερομενο ε, πρόγραμμα. Ε, ίσα ίσα θεωρώ ότι και αυτοί που προέρχονται από τον ιδιωτικό και αυτοί που προέρχονται από το δημόσιο τομέα θα πρέπει να παρακινηθούν να παρέχουν προγράμματα καλής ποιότητας και να λαμβάνουν υπόψη τους και τους θεατές τους και ακόμα και άνθρωποι σαν και εμένα είναι διατεθειμένοι να δουν προγράμματα πράγματα τα οποία μπορεί να είναι εμπορικός επιτυχή και θα πρέπει να ε, ε, παρέχονται σε ένα πολύ ευρύ και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ευχαριστώ κύριε Κύρκοφ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστώ τον Ιβο Μπέλετ. Νομίζω ότι η πρόταση έκθεση που έχουμε μπροστά μας είναι μια πολύ καλή βάση για περαιτέρω συζητήσεις όπου και κατά τη γνώμη μου χρειάζονται μόνο ορισμένε μικρέ τροποποιήσει. Γιατί νομίζω ότι καλύπτει νομίζω αναλυτικά αυτά που μα ενδιαφέρουν. Τα προβλήματα που θα πρέπει να μα απασχολήσουν, ήταν και κάποιοι συνάδελφοι σε επαφή μαζί μου γι' αυτό, είναι το θέμα κατά πόσον θέλουμε να ακολουθήσουμε την διαδικασία του κατονομάζω και <clears throat> τροπιάζω για κάποια κράτη-μέλη εγώ θα έλεγα ότι δεν πρέπει να κάνουμε, αλλά ίσως κάπως πιο γενικά να το εκφράσουμε στο κείμενο, ότι δεν ε, υπάρχουν όλοι σε αυτήν την κατηγορία. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει μια μικρή αλλαγή όσον αφορά το σημείο 6, γιατί νομίζω ότι δεν είναι καλό για μας να υπερ συγχαίρουμε την Επιτροπή για μια ανακοίνωση. Ξέρουμε ποια μορφή έχει η ανακοίνωση αυτή, αλλά ξέρω από ήμουν τότε στο Κοινοβούλιο ότι με την πρώτη μορφή της ανακοίνωσης το Κοινοβούλιο είχε μεγάλα προβλήματα. Ε, μετά έλεγαν έγιναν κάποιες αλλαγές, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο είναι σωστό η Κομισιόν με ανακοινώσει να προτρέχει νομοσχεδίων. Όχι. Λοιπόν, θα πρέπει εκεί ίσως να βελτιώσουμε την διατύπωση, γιατί στο κάτω-κάτω και μία ανακοίνωση δεν είναι τίποτα που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη. Είναι ένα πλαίσιο που δίνεται προς τα κράτη-μέλη, λέγοντάς τους εδώ θα πρέπει κάτι να κάνετε. Εκεί θα πρέπει λοιπόν στο σημείο να διορθώσουμε κάπως τη διατύπωση, κατά έχουμε μια πολύ καλή βάση Και για το άλλο θέμα θα πρέπει να δούμε πώς θα βρούμε μια καλή ισορροπία με τα προβλήματα που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη-μέλη και που προσπαθούν να ε, πολιτικοποιήσουν ή να απαγορεύσουν κατά κάποιο τρόπο τους κρατικούς, τα κριτικά μήμια ε, Πρόεδρος, και εγώ θα ήθελα να πω στον κύριο Μπελέτο ότι δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη με το σημείο 6 όπως τώρα, να μην λέμε επικροτή, να λέμε σημειώνει. Θα πρέπει όμως εδώ ταυτόχρονα να έχουμε και το θέμα που μας απασχόλησε και στην οδηγία τηλεόραση κλπ. Να πούμε δηλαδή ότι <clears throat> οι κρατικές ε, ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες είναι σημαντικές σε όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες. <clears throat> θα πρέπει κάπου να το γράψουμε αυτό. Στο 6 θα υποβάλω εγώ μια σχετική τροπολογία. Και το ίδιο ισχύει και για το ένα. Και αυτό που επίση είχε το παρατηρητήριο στο Στρασβούργο πραγματικά είχε εργαστεί πάρα πολύ καλά. Αλλιώς θα μπορούσαμε να τα διατυπώσουμε πιο θετικά. Είναι πάρα πολύ αυστηρή η διατύπωση αυτή. Έχετε εγώ έχω μια τροπολογία να υποβάλω που είναι πιο σημαντική που λέει να δώσει όλα τα απαραίτητα πόρους και ε, να ακολουθήσει την ιδέα που έχουν κατά νου τα κράτη-μέλη, να είμαστε κάπως πιο ευγενείς δηλαδή, αν θέλετε. Ωραία. Ο κύριος Μπόρις και ο κύριος Λόκεγκατ έχουν το λόγο. Ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον κύριο Μπέλετ που αναφέρεται εδώ τον αντικειμενικό χαρακτήρα των κρατικών τηλεοπτικών σταθμών. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έχουμε διαφορετικές εμπειρίες βέβαια, αλλά ακόμα και αν δούμε το παρατηρητήριο Στρασβούργο που παρατηρεί το θέμα της χρηματοδότησης των κρατικών ε, οπτικο, ε, ραδιοτηλεοπτικών ε, μέσων δεν ξέρω κατά πόσον αυτό το παρατηρείο θα μπορούσε να ασχοληθεί με το θέμα κατά πόσον τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα είναι και αντικειμενικά. Έχω ένα παράδειγμα στην Πολωνία και σε άλλες χώρες. Τα μέσα αυτά ελέγχονται από ένα πολιτικό κόμμα και ο δικός μου υποψήφιος ας πούμε παρουσιάστηκε κατά 80% αρνητικά στα ΜΜΕ. Ίσως λοιπόν αυτό το παρατηρήριο να μπορεί να ασχοληθεί και με το θέμα της αντικειμενικότητας. Το δεύτερο θέμα. Νομίζω ότι ε, τα κρατικά ΜΜΕ έχουν την υποχρέωση να ασχολούνται με την Ευρώπη και να παρουσιάσουν 180% προγράμματα που έχουν ε, προετοιμαστεί στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει, διαπραγματεύεται κάποια πρωτόκολλα με τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με τα οποία η ευρωπαϊκή παραγωγή δεν θα πρέπει να είναι στο 50% αλλά στο 35%. Είναι μεγάλη απειλή αυτή. Και μετά η Κίνα ή άλλες χώρες μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό. Και ευρωπαϊκό θα είναι μόνο το 35%. Ε, του προγράμματος που παρουσιάζεται και με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγέ μπορεί να προέρχονται και από εκτός Ευρώπης. Είναι μεγάλος κίνδυνος αυτός. Θα πρέπει να το τονίσουν. Ευχαριστώ. Πέντε ομιλητέ έχουμε ακόμα. Παρακαλώ, κανένα ένα λεπτό. Όχι να αρχίσουμε από το Α μέχρι το ΩΜΕΓΑ, αλλά μόνο αυτό που θέλουμε να συμπληρώσουμε. Κύριε Σάκα. Uh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, πολύ επικοδομητικό ο ρόλο του, για αυτό το θέμα που ενδιαφέρει πολλού. Ο εισηγητή αναγνωρίζει ότι τα δημόσια, τα ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωση είναι σημαντικά για τη δημοκρατία και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτό που είπε και ο συνάδελφο ε, Κόπ. Το δικαίωμα στην πρόσβαση σε πληροφορίες θα πρέπει να είναι δικαίωμα του πολίτη, δεν θα πρέπει να τα καθορίζει η κυβέρνηση ή ο αθέμητος ανταγωνισμός. Κάθε κράτος μέλος θα αντιμετωπίζει διαφορετικά, αλλά εγώ ενδιαφέρομαι σοβαρά για το πώς εφαρμόζουμε προδιαγραφές. Στο σημείο AIDS λέγεται ότι τα παραδοσιακά σύνορα δεν μπορούν να ισχύουν στο online περιβάλλον θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και ναι μεν όλοι λέμε ότι είναι απότομος αυτός ο δρόμος, υπάρχουν κάποια προβλήματα, υπάρχει ναι. θέμα υποψήφιων χωρών μελών, αλλά αν δεν μπορούμε να έχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο προδιαγραφών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια φιλοσοφική συζήτηση βέβαια στην οποία δεν θα ήθελα να σταθώ περισσότερο, αλλά θα ήθελα να το υπερτονίσω εδώ. Ο δημόσιος ρόλος ε, των ε, ραδιοτηλεοπτικών μέσων είναι σημαντικός, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε κίνητρα για τα καινοτομίες και να έχουμε και ε, συνεργασία μεταξύ εμπορικού και δημόσιου τομέα, γιατί πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να εξυπηρετηθούν και τα συμφέροντα του εμπορικού τομέα. Και θα ήθελα να εξετάσουμε περαιτέρω και το θέμα του ε, περιεχομένου και την ευρύτερη πρόσβαση σε μεγαλύτερο κοινό, διότι ε, ξέρω ότι θέλουμε να έχουμε πλατφόρμες για ευρύτερο περιεχόμενο και να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε μεγαλύτερο κοινό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω σαν όσα υπόθηκαν για το σημείο 12. Τη συζήτηση αυτή την κάνουν, είχαμε κάνει και για τη δική μου έκθεση περί του παρατηρητηρίου. Ο εισηγητής μίλησε για επιτήρηση των δεσμεύσεων. Δεν μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένος. Γιατί νομίζω ότι θα έπρεπε όλα αυτά να τα ορίσουμε επακριβέστατα. Τι ακριβώς θα κάνει το παρατηρητήριο, τι πληροφορίες θα μας χορηγεί να μας πείτε μερικά παραπάνω. Φερχάνη, ένα λεπτό. Θα ήθελα και εγώ καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την τόσο αναλυτική του έκδοση και τη δική σας πρόταση κυρία Πάου γιατί την ότι κινείται του προσωστή κατεύθυνση. Ακριβώς το θέμα που έδειξε μόλις τώρα ο κύριος Λόκεγκάρτ. Το παρατηρητήριο αυτό τι παρατηρεί εγώ τη θέση προ τον κύριο Μπόρις, ε, Θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνεται ο έλεγχος χωρίς να ελέγχεται το περιεχόμενο. Γιατί αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι κατά πόσον δίνεται η δυνατότητα ε, της ε, πολυμορφίας και το κατά πόσο ένα κρατικό σταθμό εκπέμπει αντικειμενικά ή όχι είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί μέσα στα πλαίσια του κρατικού εκάστοτε δικαίου. Δεν είμαστε εμείς οι Ευρωπαίοι που θα ορίσουμε τι είναι αντικειμενικό και τι δεν είναι αντικειμενικό. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται στο περιττήριο. Ευχαριστώ κύριε Καμερέβερτ. Ναι, συμφωνώ. Ήμουν πολύ ευγνώμη προ τον κύριο Πελετ που εξήγησε πώ πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτή την ε, παράγραφο ότι ακριβώς δεν πρόκειται για τον έλεγχο του περιεχομένου αλλά του ελέγχου το κατά πόσων τα κράτη-μέλη πληρούν τι υποχρεώσει τους έναντι των ε, δημοσίων, δηλαδή τηλεοπτικών σταθμών. Ε, εάν ε, ελέγχουμε το περιεχόμενο, εγώ θα είμαι αντίθετη και αυτό είναι ένας λόγος για τον οποίο καταψήφισα χθε την έκθεση Λόκεργα, δυστυχώ. Δεν ξέρω, θες να κάνει μια διευκρίνηση, ίσως λίγο έτσι τα είχα καταλάβει τα πράγματα. Ευχαριστώ τελευταίο ο κύριο Στογιάννοφ. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η έκθεση είναι πολύ καλή και συγχαίρω τον εισηγητή. Στον καιρό που μας μένει μέχρι το τέλος του μηνός θα ήθελα να προσέξουμε ιδιαίτερα το θέμα της ιότητας, όχι της ισότητας μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης. Μόνο έτσι μπορούμε να εγγυηθούμε τη δημοκρατία και τον πιλουραλισμό. Και υπάρχει και απόδειξη τούτου ότι το 2009 περίπου 200 ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί χρεοκόπησαν, πράγμα που σημαίνει ότι περίπου 2.000 νεαροί μάλλον δημοσιογράφοι βγήκαν στην ανεργία. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε εδώ τη συζήτηση. Ήβο, α όχι, έχουμε και την Κομισιόν. Ο κύριος Ζολή, ένα λεπτό και εσείς παρακαλώ. Oui, allez-y. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Entschuldigung. Ähm, le projet de rapport. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η σχέδια έκθεση μα φαίνεται ισορροπημένο, γιατί στηρίζει ένα διαδικό σύστημα. Δηλαδή, οι εμπορικοί και δημόσιοι σταθμοί μπορούν να συνυπάρξουν. Αυτό μας αρέσει. Επίσης, και εμείς συμφωνούμε ότι υπάρχει ρόλος για, τους, για τα δημόσια μέσα ενημέρωσης. Και, και ότι μπορούν και πρέπει να διατηρηθούν οι χρηματοδοτήσεις τους, όχι όμως με μοναδικό πόρο τις κρατικές επιχορηγήσεις αλλά και με άλλους. Το μόνο σημείο όπου η Κομισιόν έχει αντιρρήσεις και αμφιβολίες και το είχαμε πει και την 1η Ιουνίου η αφορά την εντολή που θα δοθεί ακριβώς στο παρατηρητήριο για την επιτήρηση του τρόπου με τον οποίο τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης γιατί έχουμε αμφιβολίες. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δικαιοδοσίες σε αυτό το τομέα σύμφωνα με το πρωτόκολλο 29 λεγόμενο πρωτόκολλο του Αμστελοδάμου και που αφορούσε συγκεκριμένα και αποκλειστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, διότι τα πρότυπα των οποίων θα επιτηρείται η εφαρμογή είναι πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτον και πρακτικότερον η Κομισιόν δεν μπορεί να χορηγήσει τέτοια εντολή χωρίς βάση του καταστατικού του παρατηρητηρίου τη συμφωνία των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος για το σημείο 12 Έχουμε αντιρρήσεις και για τους λόγους που είπαμε την 1η Ιουνίου και για κίνους που επαναλάβαμε γραπτός σε επιστολή προς τον εισηγητή. Η κυρία Λίτσα. Όχι, Ήβο, εσύ, το λόγο. παρακαλώ, σύντομα, εσύ το Ευχαριστώ πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. θα απαντήσω. Προσπάθησα να υπάρχει μια ισορροπία και να λάβω υπόψη το γεγονός ότι ε, και οι δύο πλευρές έχουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το διτό σύστημα. Ζούμε και χαλεπούς καιρούς και ο ρόλος των ιδιωτικών ε, τηλεοπτικών δικτύων και του τύπου είναι πολύ σημαντικός. Ως προς τον καταγερματισμό που ανέφερε ο κύριος ε, Κόικοπ. Υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να περιοριστούν οι επιλογές μας. Αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Ε, όπως σωστά επισήμανε η συνάδελφος, η πτυχή της επικουρικότητας ισχύει και για τη, τις χώρες και θα πρέπει να το έχουμε κατά νου και σε αυτή την περίπτωση. Ίσως θα πρέπει να έχουμε και μία παράγραφο ακόμα για το γεγονός ότι είναι ανεπαρκής η χρηματοδότηση σε κάποια κράτη-μέλη. Παράγραφος 6. Πράγματι είναι ίσως είναι υπερβολικά αισιόδοξο το θέμα αυτό και θα μπορούσαμε να το αλλάξουμε για να υποδείξουμε καλύτερα ε, τις προσδοκίες μας. Δεν μπορούμε να έχουμε αποτελέσμα τον Ιούλιο του 2009. Ε, κύριε Πάκ, τώρα, οι δικές σας παρατηρήσεις. Okay. Για την πολυφωνία και τις πτυχές αυτές. Βρισκόμαστε εν μέρη στην παράγραφο 5, αλλά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και κάτι και στην παράγραφο που μου υποδέξετε εσείς. Ε, ουσιαστικά, όμως, νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο μήκο κύματος. Ε, κύριε Μπόρης, νομίζω ότι ήταν μία από τις καλύτερες ε, κατευθύνσεις, όπως είπε και η κυρία Κάμαχερ. Τέλος, αυτή η διάσημη παράγραφος 9 για το παρατηρητήριο. Ε, άκουσα πολλές προτάσεις ε, για την παράγραφο αυτή, να τη διευκρινίσω, να τη βελτιώσω. Θα ήθελα κυρίως να διευκρινίσω εδώ, όχι όμως ως προς την εποπτεία του περιεχομένου, δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Δεν θα πρέπει να αποστείλουμε λανθασμένο μήνυμα εδώ. μας ενδιαφέρει ε, το θέμα του παρατηρητηρίου όχι μόνο από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και από πλευράς κρατών μελών να δούμε τα θέματα της ανεξαρτησίας, της χρηματοδότησης ή της ε, ελλειπούς χρηματοδότησης. υπάρχουν κάποιες πτυχές με τις οποίες συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μεν ήπια η παράγραφος, αλλά θέλει απλώς να πει ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτηματικά. Ε, Στην παράγραφο 9, να σας μεθυμίσω εδώ ένα παράρτημα το οποίο δεν το έχουμε στο κείμενο όπως διανεμήθηκε σήμερα. Ε, υπάρχει ένα άλλο έγγραφο που έχει αυτό το παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει τα, τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και εκεί διευκρινίζεται πολύ καλύτερα ε, ποια είναι τα καθήκοντα του παρατηρητηρίου. Είμαι βέβαια στη διάθεσή σας, ε, λαμβάνω υπόψη μου όλες τις προτάσεις, ε, διότι θεωρώ ότι είναι πολύ καλές. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, συγχωρέστε που είμαι μια φορά πολύ αυστηρή, αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένη που τηρήσαμε τον χρόνο μας. Λοιπόν, όποιος έχει να υποβάλει κάποια τροπολογία θα πρέπει να το κάνει μέχρι την 1η Ιουλίου, 12 το μεσημέρι. 1η Ιουλίου, 12 το μεσημέρι. Το ακούσατε όλοι. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω. Οι συντονιστές είχαν συνεδρία σήμερα το πρωί. Υπάρχουν οι αποφάσεις τους ε, στον υπολογιστή σας. Αν έχετε κάτι να επικρίνετε, σήμερα το απόγευμα στις 3. Και μην με αφήσετε μόνοι μου σήμερα το απόγευμα στις 3. Γιατί και εγώ θέλω να πάω σπίτι μου, αλλά είμαι αναγκασμένο να μείνω εδώ. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε εδώ. Ευχαριστώ και